So, gentlemen, dear colleagues, let's start. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε την ημερίδα για την εμπορική πολιτική που είναι διαρκείας μισής ημέρας, πολύ ενδιαφέρουσα για το μέλλον της εμπορικής πολιτικής. Έχουμε μια νέα επιτροπή καινούργια γενική διεύθυνση στην ε, Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και ένα νέο κοινοβούλιο και νέα διευθύντρια στην Digitrade και πρέπει να καθορίσουμε τις προτεραιότητες μας για την επόμενη πενταετία. Οπότε είχε έρθει η στιγμή να κάνουμε μια σχετική συζήτηση. Ελπίζω να είναι ζωηρή αυτή η συζήτηση. Έχουμε εμπειρογνώμονες φυσικά από διάφορους τομείς και συντονιστές, οπότε δεν θα διευθύνω τη συζήτηση εγώ μόνο ως βαρετός ο πρόεδρος Επιτροπής. Θα είναι πιο ζωντανή η συζήτηση. Θα πειραματιστούμε και με διαφορετικούς συντονιστές λοιπόν. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν θα καλήσουμε την Σαμπίν ε, Βάιαντ, Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διευθύνσης Εμπορίου, για να μας δώσει τη δική της οπτική γωνία για τις προτεραιότητες των επόμενων πέντε ετών. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η επισκόπηση δεν θα μοιάζει με την ομιλία του κυρίου Τραμπ που άκουσα χθε. Όλος ο πλανήτης συζητά περί βιωσιμότητας προκλήσεων και ένας άντρας μόνος λέει τα αντίθετα στον Ταβός. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει, αλλά και αυτό σίγουρα θα συμπεριληφθεί στην επισκόπηση που θα μας προσφέρει η Σαμπίν. Βιωσιμότητα λοιπόν, το θέμα της επιβολής και της υλοποίησης ε, της ε, εμπορικής πολιτικής επίσης μπορεί να αποδεχθούν σημαντικά στοιχεία οι εμπορικές προτιμήσεις και η σαφής αναφορά στις υποχρεώσεις ε, που ενέχουν οι εμπορικές συμφωνίες γενικότερα και πώς αυτές εφαρμόζονται και επιβάλλονται και φυσικά υπάρχουν και άλλα στοιχεία της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής που πρέπει να δείχνουν συνοχή. Ε, επίσης το ζήτημα της προσέγγισης, ε, της μηματικής προσέγγισης των διαφορών πολιτικών πρέπει να είναι και πια στο παρελθόν. Δίνω λοιπόν το λόγο στην Σαμπίν για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που οργανώσατε αυτή την εμερίδα για την εμπορική πολιτική. Δεν θα σας επικρίνω φυσικά που είναι μισή μέρα, γιατί το πρώτο μισό της ημέρας πιστεύω το αξιοποίησατε πλήρως, εγκρίνοντας με πολύ πιστική πλειοψηφία την Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών με το Βιετνάμ και τη Συμφωνία Προστασίας των Επενδύσεων επίσης με το Βιετνάμ, κάτι που πιστεύω συμβάλλει ε, στις εργασίες της δικής σας Επιτροπής. Ε, το Βιετνάμ έτσι θα είναι τέρος μα σε διάφορα ζητήματα και έχει αναλάβει τις σχετικές δεσμεύσει που θέλαμε κι εμεί. Οπότε πιστεύω η αφετηρία αυτή είναι πολύ καλή. Κοιτώντα προ το έτος που ακολουθεί, θα είναι δύσκολο για την εμπορική πολιτική. Και η περσινή χρονιά ήταν δύσκολη, το 2020 δεν θα είναι ευκολότερο. Α είμαστε ρεαλιστέ. Ταυτόχρονα, επειδή είναι πολλέ οι προκλήσει, ε, έχουμε την έναρξη μια νέα επιτροπής, το πρώτο νέο έτο ενός νέου κοινοβουλίου, νέα εντολή, νέα θητεία. Όλα αυτά αποτελούν ευκαιρία για να κάνουμε κάποιες ε, διορθώσεις ε, και προσαρμογές στι προτεραιότητές μας. Και πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε εδώ. Έχουμε ένα σημαντικό έτος μπροστά μας λοιπόν, το οποίο αναμφίβολα θα χαρακτηριστεί από αυτό που θα ονόμαζα εγώ τη μάχη ΙΠΑ και Κίνας για τεχνολογική, οικονομική και ίσως ε, στο απότερο μέλλον πολιτική ε, κυριαρχία. Επίσης φέτος θα αποχωρήσει και το Ηνωμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι πρέπει να θέσουμε τα θεμέλια για τη μελλοντική μας σχέση. Είναι εκλογική χρονιά για τη ΣΥΠΑ και επίση, φέτο ε, θα γίνουν και οι προτάσει για την Πράσινη Συμφωνία και την ψηφιακή στρατηγική. Η Κομισιόν θα υποβάλει προτάσει για αλλαγές που θα αποδειχθούν ε, ε, σημαντικές, θα μεταμορφώσουν σημαντικά τον τρόπο που ζούμε και τον τρόπο που κάνουμε εμπόριο. Οι επιδράσεις λοιπόν πάνω μας θα είναι τεράστιε. Είναι σημαντικό λοιπόν έτο το 2020, έχουμε να κάνουμε πολλά και το περιβάλλον δεν είναι δεν μας διευκολύνει την κατάσταση. Έχουμε μεγάλη πίεση στο πολυμερές εμπορικό σύστημα. Με διάφορο... Έχουμε τώρα το μηχανισμό επίλυσης διαφορών, αλλά οι εμπορικές εντάσεις δεν φαίνεται να χαλαρώνουν. Ο προστατευτισμός ε, εντείνεται όλο και περισσότερο μετά από την οικονομική κρίση. Και κοιτώντα ε, στη βάση δεδομένων μας για την πρόσβαση στις αγορές και τα εμπόδια που υπάρχουν, οι μισές καταχωρήσεις είναι από το 2015. Και ενώ όλοι παρακολουθούμε τη ΣΥΠΑ και την Κίνα, υπάρχουν και άλλε χώρε που καταφεύγουν όλο και περισσότερο στον προστατευτισμό. Η Μπέτι Τέβε ε, στο ε, κλασικό ε, κινηματογραφικό έργο All About Eve είχε πει προσδεθείτε θα είναι δύσκολη η διαδρομή. Ωστόσο, πρέπει να επανέσουμε και του εαυτού μα, γιατί έχουμε κάνει πολλά στην εμπορική πολιτική τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ένα στιβαρό θεμέλιο, ε, συμφωνίες που συνάφθηκαν, 15 μόλι την περασμένη θητεία. Έχουμε συνολικά 40 συμφωνίε που καλύπτουν περίπου πάνω από 70 χώρε. Είναι ακόμα πρόημο για να πούμε κάποια πράγματα για αυτέ τις συμφωνίε, αλλά τα σημάδια είναι καλά. Α δούμε τον Καναδά, για παράδειγμα, όπου οι εξαγωγέ μα ανέρχονται σε 41 δισεκατομμύρια ευρώ το 2018. 15% αύξηση σε σχέση με το μέσο όρο τη προηγούμενη τριετία. Είναι πολύ σημαντικό αν το συγκρίνεται με το γεγονό ότι οι εξαγωγέ προ άλλε χώρε αυξήθηκαν κατά μόλι 8%. Από μόνη τη η Γεωργία έχει αυξηθεί κατά 7%. Ε, συχνά ακούμε μόνο για τα ότι μας συμφέρει να προστατεύσουμε τη γεωργία μας και ξεχνάμε ε, τι γίνεται όσον αφορά τα συμφέροντά μας ως εξαγωγής όχι μόνο εισαγωγής. Ε, επίσης ε, έχουμε και άλλες ε, αυξήσεις πολύ σημαντικές και στην Ιαπωνία έχουμε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Είναι ακόμα νωρίς βέβαια, αλλά εδώ άρουμε σιγά σιγά εμπόδια που θα προσθέσουν 33 εκατομμύρια στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2025. Δεν είναι μόνο νούμερα όλα αυτά. Πίσω από αυτά τα νούμερα κρύβεται πραγματική ανάπτυξη και πραγματικές θέσεις εργασίας. Σήμερα η ανάπτυξη οι εξαγωγέ υποστηρίζουν 36 εκατομμύρια θέσει εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό μα συνδέει και με την παγκόσμια ανάπτυξη σε εποχέ που είναι απαραίτητη. Δεδομένου ότι τα επόμενα χρόνια το 85% τη παγκόσμια ανάπτυξη θα λαμβάνει χώρα εκτό Ευρώπη. Η εμπορική πολιτική λοιπόν φέρνει σταθερότητα και προβλεψιμότητα σε όλου του οικονομικού φορεί τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανοίγει ευκαιρίε για τι επιχειρήσει να συνεχίσουν να ε, ανθούν ε, και οι παγκόσμιες τιμές αυξάνουν ε, την ποιότητα για τους καταναλωτές. Αυτό είναι κρίσιμο και για τις μικρότερες επιχειρήσεις που βασίζονται σε τέτοιες ευκαιρίες. Οι μεγάλες επιχειρήσεις διέρχονται από αβέβαιες εποχές πιο εύκολα, αλλά για τις μικρές επιχειρήσεις υπάρχουν περισσότερες δυσκολίες και υπάρχει κίνδυνος να συνθλιβούν στο παγκόσμιο περιβάλλον. μπορούμε να δούμε και άλλα πλεονεκτήματα, αλλά να σας πω κάτι τελευταίο για το Βιετνάμ. Είναι εξαιρετική η συμφωνία. Μας δίνει πάτημα στην περιοχή ΑΖΕΑΝ, ενισχύει την παρουσία μας στην Ασία και τις δυνατότητες που έχουμε να ενθαρρύνουμε την βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή αυτή. Είναι, πιστεύω, λοιπόν, πολύ σημαντική η συμφωνία αυτή και χαίρομαι που το κοινό γενικότερα ε, επιδοκιμάζει τις πρόοδους στην εμπορική πολιτική, τις νέες συμφωνίες, τη διαφάνεια ε, που έφερε στην εμπορική πολιτική η παλιά ε, επιτροπή. Όλα αυτά αναγνωρίζονται και υπάρχει ευρύτερη δημόσια υποστήριξη για την εμπορική πολιτική, κάτι στο οποίο θα πρέπει να βασιστούμε για το όσα θα κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Να σας πω τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Μιλάμε για το εμπόριο. Και όταν μιλάμε για εμπόριο σήμερα δεν μιλάμε πάντα μόνο για εμπορική πολιτική. Το εμπόριο χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο μιας άλλης, ενός άλλου θέματος του της μάχης για τεχνολογική κυριαρχία και για αυτήν χρησιμοποιείται το εργαλείο το εμπόριο. Περιλαμβάνει την τεχνολογία, την ασφάλεια, ε, τα οικονομικά. Είναι μια πρόκληση στην οποία πρέπει να προσαρμοστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών δεν βοηθά ε, σε αυτή την προσαρμογή σίγουρα, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Τόσο η ΕΠΑ όσο και η Κίνα επιδιώκουν μια ε, γεωγραφική και οικονομική προσέγγιση χρησιμοποιώντας τα διάφορα εργαλεία για να επιτύχουν τους στόχους. Αλλά ας είμαστε σαφείς. Πολλές από αυτές τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο πολυμερές εμπορικό σύστημα προέρχονται στην, από την ανεπαρκή ένταξη της Κίνας στην παγκοσμία τάξη. Η Κίνα έχει υποσχεθεί πολλές φορές μεταρρυθμίσεις, ωστόσο δεν έχουν γίνει ποτέ αυτές πραγματικότητα. Αν συγκρίνω τη σημερινή κατάσταση στις προσδοκίες που υπήρχαν όταν η Κίνα έγινε μέλος του ΠΟΕ το 2001, παρατηρούμε ότι οι προσδοκίες εκείνης της εποχής δεν έγιναν πραγματικότητα. Η ΕΠΑ αντέδρασαν σε αυτές τις προκλήσεις, στις ε, στρεβλώσεις ε, ε, που επιβάλλει η Κίνα ε, με αυτό το κρατικό καπιταλιστικό σύστημα. Ε, η βασική παράπλευρη ζημία αυτής της αντιπαράθεσης ήταν στον ΠΟΕ. Ο ΠΟΕ είναι ένα σύστημα που έχει υποστηρίξει τη δική μας ευημερία και ανάπτυξη εδώ και δεκαετίες θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε το βιβλίο κανόνων του ΠΟΕ ώστε να αντιστοιχεί στις προκλήσεις του 21ου αιώνα και να μπορεί να αντιμετωπίσει μια χώρα του, μεγέθους, ε, του οικονομικού μεγέθους της Κίνας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε κάποιες διορθώσεις στο σύστημα και αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα για αυτή την Επιτροπή. Αλλά φυσικά το εμπόριο δεν υπάρχει μόνο του πρέπει να συμβάλλει και σε άλλους τομείς πολιτικής επίσης και το κεντρικό κομμάτι στο οποίο θα ήθελα να εστιαστώ γιατί δεν θα είμαι εδώ για τη συζήτηση του πάνελ για τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά θέλω να το αναφέρουμε πρέπει να δούμε πώς το εμπόριο συμβάλλει στην Πράσινη Συμφωνία πώς μπορεί να συμβάλλει στην Πράσινη Συμφωνία καταρχάς πρέπει να διαβεβαιωθούμε ότι η εμπορική πολιτική δεν προκαλεί ζημίες ή βλάβες αυτός είναι ο βασικός κανόνας το να μην προκαλείς βλάβες αλλά αυτό χρειάζεται, σημαίνει ότι χρειάζεται να αλλάξουμε ελαφρώ και τη θέση μα, να την προσαρμόσουμε περισσότερο. Εμπόριο σημαίνει περισσότερε μεταφορέ, περισσότερε φιλοδοξίε και περισσότερε εκπομπέ, εκπομπέ που είναι κακέ για το, περιβάλλον. Ωστόσο αυτή η αξιολόγηση είναι απλή. Πρέπει να αξιολογήσουμε πλήρω τι εμπορικέ μα συμφωνίε και τι εμπορικέ μα ροέ και να δούμε τι επιρροή έχουν για το περιβάλλον και για το κλίμα. Είναι καλύτερα για το κλίμα το να αγοράζει κανεί ουσιαστικά φράουλε οι ντομάτες από το Μαρόκο παρά να ε, τις καλλιεργεί σε θερμοκήπια στη Βόρεια Ευρώπη. Αλλά αυτό είναι ένα παράδειγμα. Τα πουλερικά από τη Βραζιλία και τη Νέα Ζηλανδία ε, έχουν υψηλές εκπομπές. Αλλά όλα αυτά πρέπει να τα δούμε με τις σχετικές αξιολογήσεις και τις εκτιμήσεις. Αλλά δεν, είμαστε, δεν σταματάνε εκεί οι φιλοδοξίες μας. Πρέπει να δούμε πώς το εμπόριο θα μπορούσε να συμβάλλει θετικά για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενθαρρύνοντας την καινοτομία, ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις ε, σε παραγωγή ε, χαμηλού άνθρακα, ε, στην παραγωγή περιβαλλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών. Όλα αυτά πρέπει να τα ενισχύσουμε πολυμερώς και στις διμερείς μας σχέσεις. Και τρίτον, υπάρχουν τομείς όπου τα εμπορικά μέτρα ενδέχεται να αποδειχθούν αναγκαία, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της κλιματικής μας πολιτικής. Εκεί ε, επισέρχεται ο μηχανισμός ε, προσαρμογής του άνθρακα στα σύνορα, διότι μόνο αυτό θα δώσει ε, την βεβαιότητα στα κράτη και στις επιχειρήσεις της Ευρώπης για να αυξήσουν τις φιλοδοξίες τους για μείωση των εκπομπών. Αν μπορούμε να τους διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε οποιοδήποτε πειρασμό για μετακίνηση τη παραγωγή εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπιστεί από εμά. Ε, γιατί κάτι τέτοιο θα έχει ω αποτέλεσμα να ξαναμπαίνουν στην Ευρώπη προϊόντα που ρηπαίνουν περισσότερο. Οπότε θα δούμε του τομεί ε, που υπάρχει υψηλό κίνδυνο διαρροή άνθρακα και θα αξιολογήσουμε τα καλύτερα μέτρα που υπάρχουν. Θα γίνεται δηλαδή μια εκτίμηση αντικτύπου στην οποία θα συμμετέχει και το Κοινοβούλιο. Η Κίνα, ωστόσο, θα πρέπει να παίξει ρόλο και σε, παίζει ρόλο και σε άλλου τομεί όπου πρέπει να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μα. Ανέφερα ήδη την εμπορική ασφάλεια και την τεχνολογία. Αυτό σχετίζεται με ολόκληρη τη στρατηγική μα στο πλαίσιο τη εμπορική πολιτική. Το ζήτημα τη τεχνολογική κυριαρχία είναι σημαντικό. Θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση για το ποιοι είναι οι κλάδε όπου δεν έχουμε περιθώριο να εξαρτώμαστε από παραγωγέ εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιε είναι οι βασικέ τεχνολογίε, τεχνολογίε κλειδιά που χρειάζεται να έχουμε εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται να έχουμε ασφαλεί αλυσίδε προμηθειών, υψηλή προστασία τη διανοητική ιδιοκτησία, ενώ θα τηρούμε ταυτόχρονα και του κανόνε τη ελεύθερη αγορά και του ανταγωνισμού. Ήδη εργαζόμαστε σε αυτό τον κλάδο με τον έλεγχο των επενδύσεων και τη μεταρρύθμιση του κανονισμού για τα προϊόντα διπλής χρήσης. Ωστόσο, το εμπόριο θα πρέπει να συμβάλλει σε όλου του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη και χαίρομαι που αργότερα θα ασχοληθείτε αποκλειστικά με αυτό το θέμα. Έχουμε ήδη τα εργασιακά δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα περιβαλλοντικά και τα καταναλωτικά πρότυπα. Όλα αυτά έχουν συμπεριληφθεί στι ε, συμφωνίε μα και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα εφαρμοστούν. Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για μια ολοκληρωμένη και συνεκτική εμπορική πολιτική. Αλλά ήθελα να σα προειδοποιήσω μην έχετε υπερβολικέ προσδοκίε από την εμπορική πολιτική. Η εμπορική πολιτική μπορεί να συμβάλλει σε κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορεί να διορθώσει όλα τα προβλήματα που έχουμε. Η εμπορική πολιτική δεν είναι εξωτερική πολιτική, ούτε πολιτική ασφαλεία, ούτε αναπτυξιακή, ούτε κλιματική πολιτική. Το εμπόριο θα πρέπει να εστιάζεται στα αυτά που μπορεί να επιτύχει. Που, σε αυτά που κάνει καλά, φέρνει ευημερία, ενισχύει την οικονομία, είναι η ατμομηχανή ε, τη, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας τι θα κάνουμε το 2020. Είπα ήδη το να φτιάξουμε τον ΠΟΕ ε, μεταρρυθμίζοντας ε, τη διαπραγματευτική του, το διαπραγματευτικό του ρόλο και ε, για την καθιέρωση του μηχανισμού επίλυσης διαφορών. Δεύτερον, ε, διαχείριση των βασικών μας σχέσεων με τη ΣΥΠΑ και την Κίνα, όπως έγινε μια συνάντηση μεταξύ της κ. Βαντερλάιν και, και του Πρόεδρου Τραμπ στον Ταβός, για να δούμε πώς μπορούμε να ανανεώσουμε την διατλαντική σχέση. Επίσης συνεργαζόμαστε με την Κίνα. Ε, γίνονται διαπραγματεύσει για μια επενδυτική συμφωνία που θα εξετάσουν διάφορα θέματα όπως η αναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας σε κρατικές επιχειρήσεις. Επίση, αυτό σημαίνει διαφοροποίηση των σχέσεών μα. Γι' αυτό καλωσορίζουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί εδώ με το Βιετνάμ. Θα χρειαστεί να βρούμε ε, κάποιο νέο τρόπο συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τι προσπάθειε με την Ελβετία μελετάμε μια νέα στρατηγική φέτο με την Αφρική. Θα γίνει και μια σύνοδο κορυφή ε, σύντομα. Όλα αυτά είναι σημαντικά, όχι μόνο στο πλαίσιο τη εμπορική πολιτική και των εμπορικών συμφωνιών. Ε, θα μα βοηθήσουν να κινηθούμε σε ένα κόσμο ε, όπου οι πολυμερεί κανόνε βρίσκονται υπό απειλή. Και φυσικά θα πρέπει να παρακολουθούμε ότι επιτυγχάνονται, ότι φέρνουν αποτελέσματα όλε αυτέ τι συμφωνίε, ότι δεν παραμένουν απλά νεκρό γράμμα, αλλά ότι θα εντάξουμε και τις δικές μας δραστηριότητες επιβολής ε, στις σχετικές υπηρεσίες, ούτως ώστε η προβλεψιμότητα να είναι μεγαλύτερη όσον αφορά τις προσπάθειες υλοποίησης. Και τέλος, η ίση ώρα ανταγωνισμού. Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον εκτό εμπόριο, αλλά δεν πρέπει να είμαστε αφελείς. Ενώ πάντα θα προτιμάμε τη διαπραγμάτευση είτε διμερή είτε πολυμερή, θα πρέπει να μπορούμε και να αμυνθούμε όταν ε, οι άλλοι δεν θέλουν να διαπραγματευτούν μαζί μας. Πρέπει λοιπόν να προστατευόμαστε από τις αθέμητες πρακτικές. Γι' αυτό το λόγο θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία υπεράσπισης του εμπορίου ανάλογα με το πώς ε, χρειάζεται και έχουμε κάνει και μια πρόταση για τη μεταρρύθμιση του κανονισμού επιβολής. ούτως ώστε να χρησιμοποιείται και το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ. Ε, θα πρέπει να δούμε και το εργαλείο των δημοσίων συμβάσεων και ε, στην Επιτροπή επίσης ασχολούμαστε με τις διαστρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά λόγω των ξένων επιχορηγήσεων. Για όλα αυτά τα ζητήματα, για όλο αυτό το θεματολόγιο, χρειαζόμαστε ισχυρή συνεργασία μεταξύ Κομισιών, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη κοινωνία των πολιτών. Υπό όλε τι μορφέ. Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο τόσο για την αποτελεσματικότητα όσο και για την ομιμότητα τη εμπορική πολιτική. Οι πολίτε έχουν εύλογα ερωτήματα για την εμπορική πολιτική και πιστεύω δεν θα καταφέρουμε να τα απαντήσουμε μόνοι μα στην Κομισιόν. Χρειαζόμαστε μια ενημερωμένη συζήτηση πιστεύω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το καταλληλότερο μέρο για μια τέτοια συζήτηση. Αλλά αυτή η συζήτηση πρέπει να μεταφερθεί και στα κρατημέλη και σε τοπικό επίπεδο, διότι σε τελική ανάλυση, όπω σε όλε τι πολιτικέ και η εμπορική πολιτική, είναι το ίδιο. Εδώ θα κλείσω και αναμένω τι ερωτήσει για να συνεχιστεί η συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Σαμπίνε για αυτή την ε, εικόνα που μας έδωσες για την προοπτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Διεύθυνσης Εμπορίου. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην ε, συντονίστριά μας, κυρία Ιωάννα Ντράιερ, που είναι ε, εκδότης του Bordelex, που είναι ένα ε, εσωτερική, μια εσωτερική ενημερωτική επιστολή για την εμπορική πολιτική. Ε, σας ευχαριστώ πολύ, τιμή μου που με καλέσατε και που είμαι σήμερα εδώ και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να συζητήσουμε την εμπορική πολιτική μέσα στο 2020. Ε, και εγώ πρέπει να γράψω και ένα σχετικό άρθρο στο εν λόγω έντυπο. Μιλάμε για την εμπορική πολιτική σε τεραχώδεις καιρούς. Έχουμε διάφορους ομιλητές με ε, σπουδές οικονομίας, ε, νομικές και ε, εμπορικού, εμπορικές. Η Σαμπίνε θα μείνει μαζί μας για να συζητήσουμε για την επόμενη μια μισή ώρα και μετά θα πάμε στην επόμενη πάνελ. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στους ίδιους ομιλητές. Πρώτα έχουμε Έχουμε πρώτα την Στέλιγκερ που είναι ε, αναπληρωτής γενική διευθυντής ε, στην ε, με συγχωρείτε, την κυρία Τζούλια Νίλσον που είναι αναπληρωτή διευθυντής του τμήματο ε, Μπόριο και Γεωργία του ΩΣΑ, τον Πίτα του καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του ε, Λονδίνου ε, και την Άννα Στέλιγκερ που είναι αναπληρώτρια διευθύντρια στην Ομοσπονδία στον, στον ε, βιομηχανικό σύνδεσμο της Σουηδίας. Λοιπόν, ας ακούσουμε πρώτα τη Τζούλια Νίλσον. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι σήμερα εδώ και να σας δώσω κάποιες ε, σκέψεις από τη δική μας προοπτική. Εγώ μόνο να, να την εικόνα που περιέγραψε η Σαμπίνε ε, σε σχέση με τους δύσκολους καιρούς που διανύει το εμπόριο. Και δεν είναι μόνο το τι συμβαίνει, είναι και η αβεβαιότητα για το τι θα συμβεί αργότερα, γιατί δεν ξέρουμε πια και αυτή η αβεβαιότητα βλέπουμε να έχει μεγάλο αντίκτυπο στις επενδύσεις και αυτό καθυστερεί ε, και μειώνει την παγκόσμια ανάπτυξη. Μιλάμε για διεθνή συνεργασία Α, ξέχασα να σου πω λίγο πιο αργά αν γίνεται να μιλάς και καθαρά γιατί έχουμε διερμηνείς ε, για όλες τις γλώσσες και έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο από ό,τι σκεφτήκαμε στην αρχή οπότε είμαστε εντάξει από άποψη χρόνου. Ναι, συγγνώμη που μιλάω γρήγορα λέει η ομιλήτρια η κυρία Νίλσον. Καθώς σκεφτόμαστε τις προκλήσεις λοιπόν ε, της παγκόσμιας συνεργασίας και της ε, παγκόσμιας νομοπαραγωγικής διαδικασίας, ε, αυτή η αβεβαιότητα επηρεάζει τα πάντα και είναι βλαβερή κυρίως για τις μικρές εταιρείες και πρέπει αυτό να το σκεφτούμε και όσον αφορά τον αντίκτυπό του στην παγκόσμια μεγέθυνση. Χρειαζόμαστε διεθνή συνεργασία και ε, παγκόσμιο νομοθεσία. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζει το σύστημα εμπορίου τη σήμερα ημέρα είναι αυτές που απαιτούν παγκόσμιες λύσεις και ολοκληρωμένες λύσεις. Πρώτον, ε, πρόκειται για την ψηφιοποίηση και το ψηφιακό εμπόριο που αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζει το πώς εμπορευόμαστε. Έχουμε το παγκόσμιο ίντερνετ, το οποίο όμως σκοντάφτει σε εθνικές νομοθεσίες ιδιαίτερα στο πολύ δύσκολο το θέμα των διασυνοριακών ροών δεδομένων. Και εδώ έχουμε διαφορετικά ρυθμιστικά καθεστώτα και πρέπει να βρούμε κάποιο είδους διαλειτουργικότητα, μια λύση, εάν θέλουμε να ε, ωφεληθούμε ε, από την ψηφιοποίηση για το εμπόριο για όλους, δηλαδή για μικρές εταιρείες, για τις γυναίκες, για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, Ε, υπάρχουν διαφορέ πούμε, στην προστασία δεδομένων ε, μεταξύ ήπα και Ένωση. Ε, είναι σημαντικές, αλλά πρέπει εμείς να βρούμε τρόπο αυτό το πρόβλημα να το μειώσουμε και να μην αφήσουμε να μας εμποδίσει μια τάση που επιβάλλει ευρύτερες, ευρύτερους περιορισμούς για σημαντικά μεγάλα κομμάτια δεδομένων, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες. Το γεγονός ότι υπάρχει το παγκόσμιο ίντερνετ και πρέπει να το διατηρήσουμε, θέλουμε να το διατηρήσουμε παγκόσμιο, πρέπει να μας οδηγήσει στην εξέβρεση λύσης. Δεύτερον είναι οι επιδοτήσεις, οι κρατικές ενισχύσεις στο γεωργία, στο καύσιμα και ούτε καθεξής. Τώρα βλέπουμε να γίνονται αλλαγές και να επηρεάζονται και διάφοροι βιομηχανικοί τομείς. Πρόκειται για μια βιομηχανία ανάπτυξης και οι κυβερνήσεις αισθάνονται τις εξής πιέσεις. Πρώτον ανησυχούν κατά των ε, ε, βαθιά εδρεωμένων καπιταλιστικών θυλάκων. Ε, Έπειτα φαίνεται να υπάρχει κίνηση πιο δυναμική στο ψηφιακό τομέα και τρίτον να τους ανησυχεί το να μείνουν εκτός αγορών input και output μέσα σε αυτού του είδους τις εμπορικές δραστηριότητες. Με αυτό το υπόβαθρο είναι μεγάλος ο πειρασμός να κλείσουν οι αγορές να, που, ε, να ρηχτεί δημόσιο χρήμα σε διάφορες δραστηριότητες. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο κατά τη γνώμη μας σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι στρεβλώνει τις αγορές, στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και υπάρχει κίνδυνος υπερπαραγωγικότητας Υπάρχει ο κίνδυνος για πόλεμο επιδοτήσεων που θα είναι πολύ βλαβερός ειδικά προς τις, ε, απέναντι στις αναπτυσσόμενες χώρες που δεν έχουν τόσα χρήματα στη διάθεσή τους αλλά και όσον αφορά τις ε, χώρες αγορές που δεν θέλουν να ενισχύουν ε, να επιδοτούν. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν επιτρέπεται και απαγορεύεται διαρροπάλου η επιδότηση. Μπορεί να χρειαστεί να βοηθηθούν ας πούμε, αυτοί που επηρεάζονται από την ψηφιοποίηση, αλλά συχνά οι κρατικέ ενισχύσει δεν πάνε εκεί που πρέπει, αλλά σε κλάδους που επιδοτούνται καθαρά και πολύ μόνο Δηλαδή δεν, μπορούμε παρά να λύνουμε ε, τα χτεσινά και προχτεσινά προβλήματα τα οποία σωρεύονται. Εάν θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα των επιδοτήσεων θα πρέπει να το δούμε, να δούμε τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Τώρα, η συσχέτιση μεταξύ εμπορίου και βιωσιμότητας. Εδώ χρειάζεται πηγόντως παγκόσμια συνεργασία αν θέλουμε να μειώσουμε τις ε, εκπομπές. Υπάρχουν όμως δύσκολα ζητήματα σχέσεις ε, ανάμεσα στις περιβαλλοντικές συμφωνίες και τις περιβαλλοντικές συμφωνίες και πώς μπορούν ε, αλλήλως να βοηθηθούν Υπάρχουν ε, δύσκολα και τεχνικά θέματα για να σχεδιάσουμε μέτρα ώστε να στοχεύσουμε στο, σε ένα πρόβλημα και να είμαστε αποτελεσματικοί. Και υπάρχουν και επίση και αυτά τα θέματα που αφορούν τον αντίκτυπο για την εγχώρια οικονομία και τον πληθυσμό τη κάθε χώρα. Ποιο πληρώνει και πώ. Και όταν μιλάμε για παγκόσμια συνεργασία, να πω τέλο, ε, πω συχνά αυτό έχει να κάνει με το εθνικό επίπεδο και τι εσωτερικέ πολιτικέ ιδιαίτερα σε ένα τομέα κλειδί που είναι η απώλεια δημόσιας στήριξης για το εμπόριο. Γιατί έχουμε μεγάλους αριθμούς ανθρώπων που πιστεύουν πως η παγκοσμιοποίηση δεν τους ε, βοηθά και οι εσωτερικές πολιτικές δεν είναι επαρκείς επίση. Εάν θέλουμε να προχωρήσουμε λοιπόν με την παγκοσμιοποιημένη οικονομία πρέπει να βρούμε παγκοσμιοποιημένες λύσεις. Ε, ε θα πρέπει ίσως να προωθήσουμε πράγματα ε, που θεωρούμε πως έχουν λειτουργήσει θετικά, αλλά αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αν δεν υπάρχει ψηφιοποίηση και αν βάλουμε τις ενισχύσεις σε λάθος τομείς, δεν θα έχουμε τα εργαλεία και ούτε και τους δημόσιους πόρους που χρειάζονται για να βοηθήσουμε και να αντιμετωπίσουμε σε αυτές τις πολύ δύσκολες καταστάσεις. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την εισήγηση αυτή. Μπήκατε κατευθείαν ε, στα βαθιά νερά. Πείτε πώς πάει το σύστημα, μπορείς να μας πεις. Να σας πω πώς πάει το σύστημα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να μπορέσω να απευθυνθώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ θα προσπαθήσω να μιλήσω γενικότερα, να σα δώσω μια συνολική εικόνα τη πολιτική ε, σε ζητήματα διεθνού εμπορίου, που φυσικά θα είναι ε, μια ευρύτερη παρουσίαση, μιας και έχουμε και λίγο χρόνο. Και θα σταθώ σε δύο ε, πολύ σημαντικά παράδοξα στο, στην πολιτική εμπορία αυτή τη στιγμή. Εγώ το ονομάζω παράδοξα. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει ότι πρόκειται για μια κατάσταση που δημιουργεί τριβές. Εγώ προέρχομαι από ένα κράτος μέλος το οποίο σύντομα θα εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα προσπαθήσω να μην χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, τη λέξη την κακή που ξεκινάει από B, αλλά θα αναφερθώ ακριβώς στο ζήτημα των προσκομμάτων των εμποδίων στο εμπόριο. Και, και συχνά γίνονται αυτές οι αναλογίες, οι μεταφορές σε σχέση με τους πολέμους, δηλαδή τον πόλεμο τον εμπορικό, ή το, παλιά τον πόλεμο των άστρων. Ε, η παλια τον πολεμο των αστρων η κυβερνηση Τραμπ χρησιμοποιεί τις κυρώσεις ως μέσο πίεσης για να αποσπάσει συμφωνίες και η επιβολή δασμών επανήλθε στην ημερήσια διάταξη. Και αυτό, κατά την άποψή μου, είναι ένα μεγάλο παράδοξο, γιατί το διεθνές εμπόριο κατά την άποψή μου σήμερα θα έπρεπε να ασχολείται, να, να εστιάζει πολύ περισσότερο σε ζητήματα ρυθμιστικά και συντονισμού των διαφορετικών ρυθμιστικών πλαισίων παρά να ξαναμιλούμε για δασμούς το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι ακόμα πιο σημαντικό όταν έχουμε μια παγκόσμια οικονομία αλληλοεξαρτώμενη και αλληλοσυνδεδεμένη. Πολύ πιο σημαντικό από τους δασμούς. Βεβαίως με μια εξαίρεση είναι κάτι διαφορετικό να μιλούμε για μια αναπτυσσόμενη χώρα η οποία θα χρειάζεται να βοηθηθεί και να προστατεύσει την οικονομία τη μέσω των δασμών. Θα μπορούσα να μιλώ πολύ γι' αυτό, αλλά θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, μια ομιλία χτεσινή του Διευθύνοντος Συμβούλου τους Google, η οποία, στην οποία αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξουν ρυθμίσεις για το ίντερνετ, για την ψηφιακή οικονομία. Ε, σήμερα όλοι αυτό το αντιμετωπίζουν ως ένα ζήτημα εμπορικής πολιτικής. Επίσης πιστεύω ότι υπάρχει και ένα βαθύτερο φιλοσοφικό ζήτημα, το οποίο δεν μας βοηθά να αντιληφθούμε ποια είναι τα διάφορα ζητήματα τα οποία συνδέονται με την εμπορική πολιτική. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφερόμαστε στην κοινή εμπορική πολιτική, και, αλλά αυτό δεν, κοινή οργάνωση όλα, όλα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν πλήρω τη σημερινή διεθνή πραγματικότητα, το πόσε πολλέ αλληλεπιδράσει και σχέσει υπάρχουν μεταξύ των κρατών σε εμπορικό επίπεδο. Γιατί δίνει την εντύπωση ότι η εμπορική πολιτική είναι κάτι μια μορφή εξωτερικής πολιτικής. Είναι κάτι που εφαρμόζουμε στα σύνορα, στα ε, αγαθά και τις υπηρεσίες που εξάγουμε και εισάγουμε. Βεβαίω αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο μια διεθνού εμπορική πολιτική, αλλά η διεθνή εμπορική πολιτική είναι πολύ ευρύτερη. Κατά την άποψή μου, για παράδειγμα, ο Γενικό Κανονισμό Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, που επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων, είναι εξίσου σημαντικό με άλλα στοιχεία τη εμπορική πολιτική, όπω για παράδειγμα η Τελωνιακή Ένωση. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο παράδοξο που διαπιστώνουμε στη διεθνή σκηνή. Να ξαναμιλάμε για δασμούς, ενώ στην πραγματικότητα τα ουσιαστικά ζητήματα έχουν σχέση με το ρυθμιστικό πλαίσιο. Το δεύτερο παράδοξο, κατά την άποψή μου επίσης ε, συνδέεται με το πρώτο. συνεχίζοντα την αναλογία και την αναφορά στον πόλεμο των άστρων, θα έλεγα ότι έχουμε την επίθεση κατά του πολυμερούς συστήματος διαπραγμάτευσης. Ε, γνωρίζω πόσο δύσκολο θα είναι η συζήτηση και η διαπραγμάτευση της Σαμπίν και σας εύχομαι καλή τύχη στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Αυτό συνδέεται άμεσα με το παράδοξο των δασμών. Γιατί, Γιατί κατά την άποψή μου η παγκόσμια πολιτική στα ρυθμιστικά ζητήματα δεν μπορεί παρά να προαχθεί εάν, ε, παρά μόνο μέσω πολυμερών συμφωνιών σε διεθνή φόρα. Προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, με τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου να προωθήσει τέτοιες, ε, τέτοιο συντονισμό σε ρυθμιστικό επίπεδο, αλλά εάν δει κανεί διαπραγματεύσει όπω η διαπραγμάτευση για την TTIP, η διαπραγμάτευση για τη ΣΥΤΑ, διαπιστώνει πόσο δύσκολο είναι να σημειωθεί πρόοδο σε ρυθμιστικά ζητήματα όταν αυτό γίνεται με διμερή διαπραγμάτευση. Άρα, κατά την άποψή μου, στα ζητήματα τα ρυθμιστικά δεν υπάρχει άλλη παρά μεταξύ της πολυμερούς συνεννόησης των κρατών ή των μονομερών ενεργειών. Αυτά είναι λοιπόν είναι τα δύο μεγάλα παράδοξα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και κλείνω Προσπαθώντα να περιγράψω ποια είναι, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να είναι η θέση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτά τα δύο παράδοξα και τι θα πρέπει να κάνει. Κατά την άποψή μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο σημαντικότερο οικονομικό, ρυθμιστικό παίκτη στον κόσμο. Ίσως να είναι λίγο υπερφύαλο αυτό που λέω, αλλά το πιστεύω πραγματικά. Και δεδομένου ότι προέρχομαι και από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα έλεγα ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι ε, εύλογη η πολιτική, η ρυθμιστική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο καταφέρνει να ε, κρατάει σε χαμηλό επίπεδο τις λαϊκιστικές φωνές. Είναι πολύ δύσκολο για μια, για μια ένωση όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει λαϊκιστικές εμπορικές πολιτικές στο διεθνές επίπεδο. Δεν μπορώ να φανταστώ την Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, να χρησιμοποιεί τους δασμούς όπως ο Τραμπ, ε, μπορεί βεβαίως και πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να προωθεί τα στοιχεία που κάνει, όπως για παράδειγμα τα ζητήματα τα εργατικά ή την πολυμερή, τις πολυμερείς ε, διαπραγματεύσεις. Και να προσπαθήσει να πείσει τους ηγέτες να επανέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά αυτό όχι μόνο προσπαθώντας με πειθό να εξηγήσει γιατί τα προβλήματα είναι σημαντικά και χρειάζονται συνεννόηση, αλλά επίσης αξιοποιώντα και μονομερείς ε, ε, με μνημονία επιβολή μέτρων. Δεν το έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Καταπιστεύω ότι τα επόμενα λίγα χρόνια θα χρειαστεί να το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο λοιπόν να συζητήσουμε αυτή την πρόταση που σας κάνω σε σχέση και με το επόμενο πάνελ, δηλαδή την ε, σημασία του διεθνούς εμπορίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη, γιατί αυτό είναι ένας τομέας στον οποίο πιστεύω ότι η μερομονομερής πιθανώς δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Σας ευχαριστούμε να δώσω το λόγο στην Άννα να μας δώσει και την σουηδική προσέγγιση. Ευχαριστώ και πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας τόσο επίκαιρα ζητήματα, τόσο σημαντικές συζητήσεις ε, για την εμπορική πολιτική. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν οι προηγούμενοι μιλητέ. Έχουμε ακούσει ότι ο κόσμο αλλάζει, το γεωπολιτικό πλαίσιο αλλάζει και θέλω να σα υπενθυμίσω ότι και το ίδιο το εμπόριο επίση αλλάζει. Θα ήθελα να παραθέσω κάποια πράγματα στα οποία θα θέλαμε να επικεντρωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Επειδή όλα αλλάζουν, παρότι μερικές φορές βλέπουμε φυλάδια ενημερωτικά για το εμπόριο με ε, κοντέινερ που κυκλοφορούν πάνω σε ωκεανούς ε, και μέσα από σύνορα, ξέρουμε ότι το εμπόριο σήμερα δεν αφορά μόνο την ροή εμπορευμάτων αλλά και ανθρώπων, δεδομένων, υπηρεσιών, κεφαλαίου, ιδεών, αφορά πρότυπα, αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, αφορά τις θέσεις εργασίας. Όλα αυτά σε εποχές ε, ταραγμένες. Οπότε θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για τις τεράστιες αλλαγές που έχει υποστεί το ίδιο το εμπόριο σήμερα και μετά να σας τονίσω ποιο θα μπορούσε να είναι το μέλλον της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας, δούμε, ας πάμε λίγα βήματα πίσω να δούμε τις μεγάλες αλλαγές που έχει υποστεί το εμπόριο. Τρεις θεωρώ ότι ήταν οι μεγάλες αλλαγές. Ε, οι τρεις μεγάλες αλλαγές, όπως θα μπορούσαμε να τις πούμε, οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, η ψηφιοποίηση και οι άλλες αλλαγές. Για δύο δεκαετίες μιλάμε για την παγκοσμιοποίηση. Συζητήσαμε πολύ για την παγκοσμιοποίηση, αλλά η παγκοσμιοποίηση βλέπουμε τώρα πώ έχει αλλάξει σε βάθο και πρακτικά τον τρόπο που παράγουμε, που εμπορευόμαστε και που καταναλώνουμε. Η πρώτη λοιπόν μεγάλη τάση, οι παγκόσμιε αλυσίδε αξιών είναι πραγματικότητα σήμερα, δεν είναι απλά στα λόγια. Αποτελούν πραγματικότητα για οποιαδήποτε επιχείρηση δραστηριοποιείται στο διεθνέ εμπόριο. Ξέρουμε ότι ένα φορτηγό, ένα Volvo που έχει φτιαχτεί στη Σουηδία έχει κατασκευαστεί, περιλαμβάνει πάρα πολλά χιλιάδες εξαρτήματα ε, και βασίζεται και σε υπηρεσίες παρέχονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλο και περισσότερα προϊόντα συναρμολογούνται σε μία χώρα, αλλά παράγονται σε πάρα πολλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Και η δεύτερη μεγάλη τάση πρέπει να θυμόμαστε ότι το εμπόριο είναι όλο και περισσότερο εμπόριο υπηρεσιών. Έχει αυξηθεί αυτός ο κλάδος του εμπορίου. Πάνω από το 50% του εμπορίου στις χώρες του ΩΣΑ αφορά υπηρεσίες. Αν ε, υπολογίσουμε τις υπηρεσίες αυτές, ε, χωρίς τις υπηρεσίες δεν μπορεί να υπάρξει παραγωγή. Ας δούμε μια ανεμογεννήτρια για παράδειγμα, πρέπει κάποιος να την εγκαταστήσει, κάποιος να τη συντηρεί, να την επισκευάζει, να την παρακολουθεί. Όλα αυτά γίνονται μέσω υπηρεσιών. Τρίτη μεγάλη τάση, η ψηφιοποίηση του εμπορίου, ίσως η σημαντικότερη από τις τρεις μεγάλες αυτές αλλαγές. Πάνω από το 50% όλου του εμπορίου υπηρεσιών δεν θα λάμβανε χώρα αν δεν υπήρχαν οι ψηφιακές ροές. Αν δεν υπάρχουν αυτέ οι ψηφιακέ ροέ, δεν υπάρχει λοιπόν εμπόριο. Για να πάμε στο Ινταλίκα, στο φορτηγό που σα είπα προηγουμένω, είναι σουηδική εταιρεία, δεν θα το ξανανομάσω. Σήμερα ε, πολλά πράγματα πολλούνται σε έναν πελάτη μέσω μια εφαρμογή. Έτσι έχει το εμπόριο σήμερα. Αυτέ οι τρει μεγάλε τάσει δεν είναι οι μόνε αλλαγέ που ξέρουμε. Μπορούμε να προσθέσουμε το γεωπολιτικό πλαίσιο, την αύξηση των προστατευτικών μέτρων παγκοσμίω, τι εντάσει ε, σε διαφορέ εμπορίου παγκοσμίω. Είναι σαφέ ότι η εμπορική πολιτική και το εμπορίο δεν είναι πια όπω ήταν παλιά και δεν είναι δυνατόν να είναι. Δεδομένων αυτών λοιπόν ο κόσμος του εμπορίου έχει τα τελευταία χρόνια αλλάξει σε βάθος. Ουσιαστικά μιλάμε για μια επανάσταση χάρη σε αυτές τις τρεις ε, τάσεις που ανέφερα. Να σας επισημάνω τι θα πρέπει να απασχολήσει στο μέλλον την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μου είπα να είμαι γρήγορη, οπότε από 12 στοιχεία έχω περιορίσει το κατάλογο σε 9. Κάνω ό,τι μπορώ. Απόψη ε, των επιχειρήσεων είναι σημαντικό πρώτα απ' όλα και το είπαμε, θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε τους κανόνες του εμπορίου. Ξέρουμε ότι οι παγκόσμιες ε, οι υπηρεσίε αξιών, αλυσίδες αξιών, οι υπηρεσίε και οι παγκοσμιοποίηση θα παραμείνουν, αλλά οι πολυμερεί εμπορικοί κανόνε παγκοσμίω δεν έχουν αλλάξει ανάλογα τα τελευταία 20 χρόνια. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα επικαιροποίηση των κανόνων είναι οι σημερινέ διαπραγματεύσει για το ηλεκτρονικό εμπόριο εντό του ΠΟΕ. Αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και πέρα του, ηλεκτρικού, του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι παρά ένα στοιχείο των νέων κοινών κανόνων που χρειαζόμαστε. Δεύτερο σημείο σε τραγμένες εποχές η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί να ε, υποστηρίξει ξανά και ξανά διαφανείς και προβλέψιμους κανόνες. Αυτό είναι ύψης της σημασίας για αυτούς που χρησιμοποιούν τους κανόνες, που τους ε, τηρούν, δηλαδή για τις εταιρείε. Από τέτοιους κανόνες προβλέψιμους υποφελούμαστε ε, όλοι και εκεί όπου έπαιζε κεντρικό ρόλο. Όλο λέμε ότι το πολυμερές ε, εμπορικό σύστημα ε, είναι κάτι επιθυμητό, αλλά πρέπει να το κάνουμε και δράση αυτό. Τρίτον, δεν γίνεται να γίνουν όλα στον ΠΟΕ και αυτό είναι το τρίτο μου σημείο. Πρέπει να συνεχίσουμε την φιλόδοξη ατζέντα ελεύθερων συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είχε τα τελευταία χρόνια. Και ξέρουμε ότι αυτές ε, οι συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών παρέχουν κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ καλά αποτελέσματα. Αυξάνεται το εμπόριο σε κάθε τέτοια συμφωνία κατά 50%. Και όσο πιο φιλόδοξε είναι αυτέ οι συμφωνίε, τόσο περισσότερο επηρεάζουν τα πράγματα. Τέταρτον, ε, πρέπει να είναι εύκολο για αυτού που πραγματοποιούν εμπορευματικέ συναλλαγέ να χρησιμοποιήσουν αυτέ τι συμφωνίε. Για αυτού υπάρχουν αυτέ οι συμφωνίε. Οι βελτιώσει μπορούν φυσικά να γίνουν. Χρειάζεται πιο δομημένη εμπλοκή των ενδιαφερομένων στι διαπραγματεύσει των εμπορικών συμφωνιών αλλά και στι διαπραγματεύσει εντό του ΠΟΕ όπου σίγουρα υπάρχει περιθώριο για κάποια βελτίωση. Στην MC12 στο Καζακστάν είναι δυνατόν να έχουμε κάποια επιτυχία χωρίς εμπλοκή των επιχειρήσεων, δεν είμαι βέβαιη. Πέμπτον, η ατζέντα βιωσιμότητας. Είναι αδύνατο να μην αναφερθεί θα πρέπει να εστιαστούμε και σε όλες τις διαστάσεις της βιωσιμότητας. Η εμπορική πολιτική μπορεί και πρέπει να συμβάλλει Μπορούμε να συμβάλλουμε μέσω των πολυμερών διαπραγματεύσεων στον ΠΟΕ, μέσω πολυμερών διαπραγματεύσεων, όπου δυστυχώς η Συμφωνία για τα Περιβαλλοντικά Αγαθά φαίνεται να έχει κολλήσει αυτή τη στιγμή. Μπορούμε επίσης να εστιαστούμε με τα κεφάλαια TST της Συμφωνίας Ελευθερών Συναλλαγών και μέσω των βοηθειών προς το εμπόριο η εστίαση στη βιωσιμότητα θα παραμείνει και όπως και το εμπόριο έχει συμβάλει ε, στην καταπολέμηση της φτώχειας στο παρελθόν, οπότε πρέπει να συμβάλει και στην ε, βιώσιμη ανάπτυξη στο μέλλον. Έκτον θα είμαι σύντομη. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι χρειαζόμαστε τη σχέση με τη ΣΥΠΑ. Το είπε σωστά ο κ. Χόγκαν. Πρόσφατα πρέπει να συνεργαστούμε, είπα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να σφυριλατήσουμε κανόνε εμπορικού αντί να τσακωνόμαστε για τα αυτοκίνητα και το χάλιβα. Αυτό νομίζω είπε. Ξέρω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε καλά αποτελέσματα από αυτό. Η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση, είπα και η Ιαπωνία είναι η απόδειξη. Έβδομο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποφύγει την τον βραχυπρόθεσμο πειρασμό των ωφελών των προστατευτικών μέτρων Όλοι χάνουμε σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από προστατευτισμό. Κανεί δεν κερδίζει. Ε, οι διαφανεί αξιόπιστοι κανόνε που είναι υποφελεί για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει και τι μεγάλε επιχειρήσει, τι αναπτυσσόμενες ε, χώρε και τις μεγάλες οικονομίες εξίσου, πρέπει να είναι ο στόχο λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει αξιόπιστη εμπορική φωνή προς όφελος του εμπορίου 8 υπάρχουν ε, ζητήματα γεωπολιτικά και ζητήματα ασφαλεία, Το είπαν και οι προηγούμενοι όλο και περισσότερο τίθεται ε, ε, θέμα εθνικής ασφάλειας. Οι συζητήσεις για το 5G είναι ένα παράδειγμα. Πρέπει φυσικά να αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα οποιοδήποτε ζήτημα ασφαλείας, αλλά δεν χρειάζεται να, να υποβαθμίζουμε τις φιλοδοξίες μας στον τομέα του εμπορίου. Τελευταίο, έχουμε μια φιλοδοξία ατζέντα για τα επόμενα χρόνια. Έχουμε μια νέα βιομηχανική στρατηγική, μια νέα ευρωπαϊκή συμφωνία. Όλα αυτά συζητώνται και δεν είναι παραμερικά παραδείγματα. Χρειάζεται να δείχνουμε συνοχή. Το να βασίζουμε μια ατζέντα σε αυτό που ονομάζουμε κυριαρχία δεν θα πρέπει να γίνεται εις βάρος του εμπορίου. Πρέπει να δείχνουμε κάποια συνοχή. Οπότε για να τελειώσω, ξέρουμε ότι το εμπόριο σήμερα χαρακτηρίζεται από ροέ, όπω είπα στην αρχή. Είναι μια συνεχή, απαραίτητη ροή αγαθών, ανθρώπων, υπηρεσιών, ιδεών, δεδομένων, επενδύσεων και κεφαλαίου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν πρέπει να ε, ταράσουμε τις ε, Αλυσίδε αξιών. Χρειαζόμαστε εμπόριο όπω αυτό που μα εξυπηρέτησε και που να δημιουργεί θέσει εργασία στην Ευρώπη. Όπω είπε Σαμπίν, 36 εκατομμύρια θέσεις εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζονται στι εξαγωγέ μα. Εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Οπότε μην ξεχνάμε ότι για να πάμε προ τα μπρό. χρειαζόμαστε περισσότερο εμπόριο, επικαιροποιημένου κανόνε εμπορικού, ειδικότερα καθώ μπαίνουμε σε τραγμένε εποχέ. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι μας δώσετε μια πολύ καλή εικόνα των ζητημάτων εδώ και η συζήτηση θα είναι πολύ καλή. Πριν ε, ε, δώσω το λόγο στα μέλη Σαμπίνη, μήπως θέλετε να αντιδρέσετε στα όσα υπόθηκαν. Με εντυπωσίασε το ότι συμφωνούν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όλοι οι ομιλητές. Ε, η παρατηρήση που έχω να κάνω, και αυτό είναι κάτι με το οποίο κλείνουμε, είναι ότι δεν μπορείς να είσαι από μόνος σου πολυμερής. Πώς μπορούμε λοιπόν να κάνουμε τους υπόλοιπους να επανέλθουν σε μια πολυμερή ατζέντα ώστε ε, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να το προσπαθήσουμε αυτό και οποιαδήποτε ιδέα μπορεί να έχει κανείς είναι ευπρόσδεκτη. Πώς μπορούμε να προβάλλουμε και να τονώσουμε την ενημέρωση για τις ανάγκες ε, πολυμερούς ε, δράσεις. Ίσως κάποιος εδώ στην Επιτροπή να μπορεί να έχει κάποιες ιδέες. Προτείνω λοιπόν να, συνε... να αρχίσουμε τη συζήτηση γιατί είναι πολύ συναρπαστικά αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως ε, καλύψατε ένα μεγάλο φάσμα των προκλήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια. Οπότε ίσως μια ερώτηση για να ξεκινήσω προς τη Σαμπίνε, γιατί μιλάμε για αυτό το θέμα, για τους ταραχώδεις καιρούς, για τον τρόπο που θα προχωρήσουμε, το που βρισκόμαστε, γιατί ξέρουμε βέβαια ποιες είναι οι προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ε, και βεβαίως θα θέλαμε να υπάρξει κάποια ρύθμιση Έπειτα μία παρατήρηση για το Μερκοσούρ που είναι βεβαίως μία συμφωνία την οποία προσβλέπουμε, αλλά ξέρουμε ότι κάποιοι τομείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ε, προβλήματα, κυρίως στη Γεωργία, γι' αυτό και μας ανησυχεί η τήρηση της συμφωνίας του ε, Παρισιού Υπάρχουν όμως ε, κυβερνήσεις που λένε ότι από αυτή τη μορφή δεν θα μπορέσουν να το δεχτούν. Ο Μανουέλ Μακρόν ε, και ο κύριος Κούρτς ε, ακούμε από τη Φαλονία παρόμοια μηνύματα. Το ερώτημα είναι έχουμε κανένα χώρο ελιγμού για να προσαρμόσουμε την συμφωνία ή έχετε υπόψη σας τι ακριβώς θέλουν να αλλάξουν γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Σημείο 7. Ε, πρέπει να, να, να μην ορθώσουμε νέους φραγμούς. Ε, αυτό ήταν που αναφέρατε. Αυτός ο μηχανισμός ε, για το συνοριακό άνθρακα πιστεύετε πως ακολουθεί αυτή την κατεύθυνση. Δεν θέλω να θέσω άλλες ερωτήσεις γιατί πρέπει να έχουν χώρο και οι συνάδελφοι. Κυρία Σιμακοπούλου τώρα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάλυση. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω σε κάποια πιο πρακτικά ζητήματα και πιο βραχυπρόθεσμα, γιατί έχω την εντύπωση ότι φέτος, το 2020, ξεκινήσαμε τη νέα χρονιά, μια νέα δεκαετία, νέα επιτροπή που θα έπρεπε να είναι γεωπολιτική επιτροπή, αλλά όταν πρόκειται για εμπορικές σχέσεις, κάπως ε, περίεργες ενέργειες γίνονται. Τα βασικά λοιπόν είναι νομίζω για το 2020 η Αμερική, η Αμερικανική πολιτική, πρόκειται για εκλογική χρονιά, δεύτερον το Brexit, τι κάνουμε με το Brexit και ε, γάμα ε, η Κίνα που εκεί εμπίπτει η μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, οι διμερείς σχέσεις, ε, τα όσα κάνει ο κύριος Τραμπ με τις πρακτικές που χρησιμοποιεί κτλ. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ρεαλιστικά τι πιστεύετε μπορεί να γίνει με όλες αυτές τις παραμέτρους ώστε να κάνουμε κάποια θετικά βήματα για την Ευρώπη μέσα στο 2020. Ευχαριστώ. Κύριος Βίνκλερ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τις ε, πραγματικά συναρπαστικές ε, εισηγήσει. Όλα αλλάζουν, ο κόσμος αλλάζει, η οικονομία αλλάζει, το εμπόριο αλλάζει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλάζει επίσης. Και πιστεύω τουλάχιστον να ρωτήσετε εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου, ένας από τους στόχους μας είναι να κινηθούμε προς την ίδια την εφαρμογή εμείς να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να διευρύνουμε τις αρμοδιότητές μας, πώς μπο... βεβαίως ε, συμπληρώνοντας την DG εμπορίου, τη Γενική Διευθυνσία Εμπορίου, αλλά εν πάση περιπτώσει επιφέροντας περισσότερη διαφάνεια, νομίζω πως αυξάνουμε τη δημοκρατική νομιμότητα και αυτή είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν θα μπούμε βέβαια μέσα στις λεπτομέρειες, αλλά πραγματικά ε, είμαι περίεργος και μάλιστα όχι μόνο το Ευρωκοινοβούλιο αλλά και τα Εθνικά Κοινοβούλια που συζητούν το εμπόριο και έχουν αρμοδιότητες ε, για τις επενδύσεις. Πρέπει να συμπληρώνουν δηλαδή το Ευρωκοινοβούλιο δίνοντας συνένεση στις επενδυτικές ε, συμφωνίες που είναι μειχτής αρμοδιότητας. Πώς ε, το βλέπετε εσείς. Έχω άλλη μια παρατήρηση. Έχουμε μία τύχη και διάφορες απόψεις, γιατί είπατε ότι η δημόσια στήριξη για το εμπόριο αυξάνεται, είπατε εσείς, ενώ ακούσαμε και ότι είναι ακριβώς αντίθετη άποψη. Δεν ξέρω αν έχουμε η ε, πλειοψηφία υπέρ του εμπορίου, τότε είναι σιωπηρή η πλειοψηφία. Αν έχουμε αντιπάλους του εμπορίου, σίγουρα είναι πολύ πιο θορυβόδης ε, αυτή η μειοψηφία, αν είναι μειοψηφία. Πώς λοιπόν μπαίνουμε εδώ σε αυτό το θέμα της επικοινωνίας. Οι αντίπαλοι του εμπορίου φαίνεται να χειρίζονται καλύτερα την επικοινωνία από ότι οι υπόλοιποι και φαίνεται και αυτό να είναι πρόταση του Λευκού Οίκου. Προτάσεις. Ναι, πολύ σημαντικές ερωτήσεις. Έχουμε τρεις, τις τρεις πρώτες ερωτήσεις. Πολλοί περιμένουν, θα επανέλθουμε. Αλλά θα ακούμε τρεις-τρεις τις ερωτήσεις, γιατί έχουμε μακρύ κατάλογο θεμάτων. Ποιος θέλει πρώτος να πάρει το λόγο για να μου απαντήσει. Σαμπίνε, maybe the questions to you. Σαμπίνε, <laughs> ας ξεκινήσουμε από εσάς, από τις δικές σας ερωτήσεις. Θα Ξεκινήσω από τα πιο συγκεκριμένα και μετά από τα πιο γενικά. Airbus Boeing. Αυτό μου θυμίζει αυτό το παλιό ανέκδοτο που έχουμε έναν δικηγόρο ο οποίος πάει στη, στο νομικό γραφείο του πατέρα του και του λέει μετά από λίγες μέρες Μπαμπά, πρέπει να είστε περήφανο γιατί κατάφερα να λύσω αυτή τη μεγάλη διαμάχη στην οποία εργαζόταν το νομικό μα γραφείο εδώ και χρόνια. Και του λέει ο πατέρα του: Μα τι πήγε και έκανε, από αυτού βγάζαμε λεφτά τόσο χρόνια. Αυτή είναι η περίπτωση τη Airbus και τη Boeing όπου επί 15 χρόνια πολλοί δικηγόροι και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού έκαναν μια περιουσία με αυτή τη δυναμική διαμάχη και ήρθε η στιγμή να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου για να επιληθεί αυτή η διαμάχη. Έχουμε υποβάλει προτάσεις προς τις ΗΠΑ για τα υπολοιπόμενα ζητήματα συμμόρφωσης, τα οποία, ε, στα οποία έχει καταλήξει ο ΠΟΕ με αλλεπάλληλες αποφάσεις των διαφόρων πάνελ του, επομένως είναι ξεκάθαρο ποια είναι τα ζητήματα στο τραπέζι και για αυτά έχουμε υποβάλει προτάσεις και έχουμε ζητήσει από τις ΗΠΑ να ανταποκριθούν. Μας απαντούν ότι το επεξεργάζονται, αλλά ακόμα δεν έχουμε κάποια απάντηση. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι υποβάλαμε προτάσεις για τι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο στο μέλλον θα μπορούν να δίνονται κρατικέ ενισχύσει για την κατασκευή αεροσκαφών. Γιατί δεν είμαστε μόνοι μα στον κόσμο, θα πρέπει να βρεθεί ένα γενικότερο πλαίσιο. Τώρα, σε τεχνικό επίπεδο, θα έλεγα ότι τον τελευταίο καιρό, του τελευταίου μήνε, είχαμε μια καλή ανταλλαγή με του ε, ομολόγου μα από τι ΗΠΑ. Σε πολιτικό επίπεδο, φαίνεται να υπάρχει η διάθεση να περιμένουν να δουν ε, τι θα γίνει από την πλευρά της Boeing, ε, τι θα γίνει μάλλον με την υπόθεση της Boeing και να συνεχίσουν μετά. Θα πρέπει να δούμε εάν οι Ηνωμένε Πολιτείες είναι διατεθειμένες να καταλήξουν σε κάποιο συμβιβασμό. Ε, είναι ένα ζήτημα στο οποίο δεν μπορούμε μονομερώς να επιλύσουμε. Για το Mercosur. Κατά την άποψή μου πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση θα πρέπει να ε, βασιστεί σε συγκεκριμένα στοιχεία συγκεκριμένο κείμενο και σε συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα. Ακούω πολλού να λένε με την τρέχουσα μορφή τη δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτή τη συμφωνία. Ποια είναι η τρέχουσα μορφή τη. Αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται το νομικά δεσμευτικό κείμενο. Επομένως, πριν κανείς πει ότι δεν τη δέχομαι μια συμφωνία, θα πρέπει, ή πριν κανείς να πει ότι θα πρέπει να προσαρμοστεί και να αλλάξει η συμφωνία, τουλάχιστον να ξέρουμε ποια είναι η συμφωνία ακριβώς. Ίσως το πρόβλημα να μην είναι ακριβώς το κείμενο της συμφωνίας, αλλά να είναι πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε και να υπάρξει εμπιστοσύνη της κοινή γνώμης στο ότι θα εφαρμοστεί σωστά αυτή η συμφωνία και για αυτό θα πρέπει να προετοιμαστούμε. Έχουμε χρόνο μπροστά μας, δεν ε, θα ε, κάνουμε βιαστικές κινήσεις. Θα αξιοποιήσουμε όλο το χρόνο που έχουμε για να συνεργαστούμε με τους συνεργάτες μας από την πλευρά των κρατών Μερκοσούρ για να βελτιωθούν οποιαδήποτε ζητήματα εφαρμογής. Εμείς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τη σύναψη αυτής της συμφωνίας. Νομίζω η Τζούλια, αν δεν κάνω λάθος, μίλησε για τη σχέση μεταξύ ε, συμφωνιών διεθνού εμπορίου και, και συμφωνιών για το κλίμα σε διεθνέ επίπεδο. Αυτό που κάνουμε εδώ είναι μέσω του μηχανισμού εφαρμογής μιας ε, συμφωνίας εμπορίου να τραβήξουμε τις χώρες Μερκοσούρ προς την εφαρμογή της συνθήκης των Παρισίων για το κλίμα το δείτε ε, πιο συγκεκριμένα, δηλαδή όλα τα μέτρα τα ε, ε, που δεν έχουν χαρακτήρα κυρώσεων τα οποία συμφωνήθηκαν, συνδέονται με την τήρηση της Συμφωνίας των Παρισίων. Να λοιπόν μια συγκεκριμένη προσπάθεια που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό. Το ερώτημα λοιπόν για εμένα δεν είναι τελικά το κείμενο της συμφωνίας, αλλά το πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και να διασφαλίσουμε την εφαρμογή της σωστά. Για τα αγροτικά προϊόντα έχουμε πολύ συγκεκριμένους ε, δασμούς ε, με συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλίδες ε, όλων των μορφών. Επομένως δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος εδώ αλλά αυτή η συζήτηση θα πρέπει να γίνει με ένα συγκεκριμένο νομικά δεσμευτικό κείμενο και αριθμητικά στοιχεία. Είναι μια συζήτηση που θα πρέπει προφανώ να γίνει στι Βρυξέλλε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και στο παρελθόν η Επιτροπή σα έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει περίπλοκα ζητήματα, δύσκολα ζητήματα όπω φάνηκε στην περίπτωση του Βιετνάμ. Γιατί να μην τα καταφέρουμε και για το Μερκοσούρ. για την ΑΒ, την οποία αναφερθήκατε προηγουμένω. Ε, ο Επίτροπο Χόγκαν επισκέφθηκε τι ΗΠΑ προσπαθώντα να αναθερμάνει τι διατλαντικέ σχέσει. Ε, γνωρίζω ότι θα οργανωθεί μια συνάντηση μεταξύ της Πρόεδρου Φαντελάιεν και του Πρόεδρου Τραμπ. Από τη δική μας πλευρά η πρόταση είναι ξεκάθαρη. Εμείς επιδιώκουμε και αναγνωρίζουμε τη σημασία της, του ρυθμιστικού πλησίου Θέλουμε να ε, συμφωνηθούν τα ζητήματα των δασμών, θέλουμε να ε, ε, επιληθούν οι διαφορές όχι μόνο στο ζήτημα Airbus Boeing αλλά και στο ζήτημα των δασμών στο Χάλιβα και επίσης να συζητήσουμε και το ζήτημα των πολιτικών προς τρίτες χώρες που δεν έχουν σχέση με την οργάνωση της αγοράς. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων στα θέματα αυτά και δεδομένου ότι αρνησχύουμε και εμείς τους σχετικούς μηχανισμούς δημιουργώντας ελέγχους εξαγωγών υπάρχει η διάθεση συνεργασίας με τις ΗΠΑ στα θέματα αυτά. Για το ζήτημα του Brexit. προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα το ότι, έχουμε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία πια. Έχουμε την πολιτική διακήρυξη για τη μελλοντική σχέση, έχουμε χρονοδιάγραμμα, το και πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε στα σοβαρά την ανακοίνωση που έχει κάνει η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ότι δεν, να, δεν σκοπεύει να ζητήσει επέκταση, το οποίο σημαίνει ότι με το δεδομένο χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε οτιδήποτε μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε αυτό το χρόνο και να συμφωνήσουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο ποια είναι τα ζητήματα τα κρίσιμα, στα οποία αν δεν καταφέρουμε να έχουμε συμφωνία μέχρι το τέλος της χρονιάς θα δημιουργηθούν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ε, αυτό έχει σχέση, για παράδειγμα, μάλλον ποια είναι τα ζητήματα αυτά, για παράδειγμα η συμφωνία στους δασμούς για προϊόντα, δεν ισχύει κάτι τέτοιο για τις υπηρεσίες, όσο σημαντικές και είναι οι υπηρεσίες. Το γεγονό ότι φεύγει το Ηνωμένο Βασίλειο από τις Ηνωμένες Πολιτείες από το, την κοινή αγορά, ε, σημαίνει ότι θα ξαναγυρίσουμε στο σύστημα των GATT, ε, ε, όσον αφορά το, την εμπόρια υπηρεσιών και θα δούμε αν μπορούμε από εκεί κάπως να το βελτιώσουμε στο μέλλον. Ε, είναι πολύ σημαντικό να φροντίσουμε να μην βέβαια καταλήξουμε σε μια αποχώρηση χωρίς συμφωνία να πέσουμε στο κενό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι όλα θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της χρονιάς. Εγώ πιστεύω ότι αυτέ οι διαπραγματεύσει, οι συνολικέ, θα συνεχιστούν για πολλά χρόνια ακόμα και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Για το ζήτημα της Κίνας θα πρέπει να συνεχίσουμε την εμπλοκή που έχουμε την σχέση με αυτή τη χώρα. Δεν γνωρίζω ε, να σας πω αυτή τη στιγμή αν θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε, να καταλήξουμε στη συμφωνία, της, ε, της, στη συμφωνία για την Συμφωνία Επενδύσεων μέχρι το τέλος του 2020. Παραμένουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν και πολλά ανοιχτά ζητήματα που είναι πολύ δύσκολα. Όπως για παράδειγμα το ζήτημα των, ε, ενισχύ, των κρατικών ενισχύσεω τη υπηρεσίες, τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και το ζήτημα των αναγκαστικών μεταφορών τεχνογνωσία. Ε, είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε στα σοβαρά την Κίνα ω παίκτη και θα πρέπει να φροντίσουμε, να προσαρμοστούμε, να έχουμε μια εργαλειοθήκη αυτόνομων μέτρων. Γι' αυτό, για παράδειγμα, προωθούμε τη ε, δημιουργία ενός διεθνούς μηχανισμού για τις δημοσίες προμήθειες, γι' αυτό προωθούμε μηχανισμούς ε, προστασίας της εσωτερικής αγοράς από μια επιδρομή εναντίον της από επιχειρήσεις οι οποίες θα λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις. Όλα αυτά χρειάζεται να τα προετοιμάσουμε για να φαίνεται ότι είμαστε σε θέση να κινηθούμε και αυτόνομα εάν χρειάζεται ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ενισχύει τη διαπραγματευτική μας ισχύ. Κοιτάξτε, βιαζόμαστε λίγο από χρόνο και πολλοί βουλευτές θέλουν να πάρουν το λόγο. Σας παρακαλώ κλείστε σύντομα και μετά από το δεύτερο γύρο ερωτήσεων οι υπόλοιποι μπορείτε να ενσωματώσετε τις απαντήσεις σας γιατί ο χρόνος ε, φεύγει πολύ γρήγορα. Νομίζω για την εφαρμογή νομίζω πρέπει να σχεδιάσουμε ένα σύστημα όπου θα συμμετέχουν και το κοινοβούλιο. Δηλαδή, ένα σύστημα όπου το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι κομμάτι του εγχειρήματο για το σχεδιασμό των προτεραιοτήτων και μετά να συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη και την εμπορική ε, κοινότητα. Um, Ellie Chance from the Greens who wanted to speak was on the Κυρία Chance από τους πράσινους. Δύο ερωτήσεις ήθελα να κάνω. Ε, δεν ξέρω αν θα, ποιος θα μπορέσει να απαντήσει ακριβώς. Όπως είπατε, χαίρομαι που μιλήσατε για τη σχέση του εμπορίου και της Πράσινης Συμφωνίας. Είναι σημαντική η σχέση μεταξύ των δύο και παρατήρησα ότι αναγνωρίζετε ότι το εμπόριο κάνει και παραπάνω από το απλά να μην κάνει βλάβη. Στο τέλος ομιλία σας είπατε ότι η εμπορική πολιτική δεν μπορεί να κάνει τα πάντα και αναφέρεται και διάφορα άλλα πράγματα, ευημερία, ε, δημιουργία θέσεων εργασία. Εγώ θέλω να σα πω ότι αυτή τη στιγμή αναγνωρίζουμε από κοινού ότι το εμπόριο δεν αφορά μόνο την οικονομική διάσταση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά ότι πρέπει να συμβάλλει και σε μια κοινωνική και οικολογική διάσταση. Όχι απλά να μην βλάπτει, αλλά να δρά και επικοδομητικά και δημιουργικά. Και ήθελα να σας ρωτήσω θα ζητήσετε από την DigiTrade να αναθεωρήσει όλες τις υπάρξεις εμπορικές συμφωνίες και αυτές που υποδιαπραγμάτευσε για να προσδιοριστούν πιθανέ βλάβες και πιθανή τομείς συνεργειών όπου θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τα πράγματα και όταν το κάνετε αυτό πότε θα το δημοσιεύσετε ώστε να δούμε κι εμείς πώς θα μπορούσε η εμπορική μας πολιτική να συμβάλλει στην Πρασινή Συμφωνία. Και δεύτερη μου ερώτηση αφορά τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Αναφέρατε, ε, αναφερθήκατε σε αυτό κάπως ξεχωριστά από τα υπόλοιπα θέματα, την Πρασινή Συμφωνία και την οικολογική διάσταση. Δεν μπορούμε ωστόσο να τα αντιμετωπίσουμε ξεχωριστά. Το κλίμα και τη βιοποικιλιότητα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα με το, την αποτυχία του πολυμερούς εμπορικού συστήματος. Πώς θεωρείτε ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να συνδυαστούν για να αποφύγουμε μονομερείς πρωτοβουλίες. Πώς διαχωρίζεις την επιχορήγηση ε, και την επένδυση που δεν σου αρέσει. Πώς θα κάνουμε όλα αυτά σε έναν πολυμερή τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Βόρμαν. I think all of you mentioned... Ευχαριστώ πολύ. Όλοι αναφέρατε την ψηφιοποίηση με ε, κάποιον τρόπο. Και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο και ειδικότερα για την ροή δεδομένων. Όπου όπως φαίνεται υπάρχουν πολλές διαφορετικές θέσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι είναι ζήτημα ακαιρεότητας, ε, κάτι προσωπικό, ενώ οι ΕΥΠΑ το βλέπουν ως αγαθό και εκείνα ως θέμα ασφαλείας. Τζούλια ε, Νίλσον είπε κάτι ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο τα δεδομένα το ζήτημα των δεδομένων να αποκτήσει λιγότερη σημασία και θέλω να σας ρωτήσω στο παρελ πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό τι τρόπος υπάρχει για να κάνουμε λιγότερο σημαντικό το ζήτημα των δεδομένων. Έχουμε και την κυρία Κατάιναν που θέλει να μιλήσει. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ το πανέλ για αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Ε, ήταν ιδιαίτερα πλήρες. Εμένα θα με ενδιαφέρει να καταλάβω πώς συνδέεται το παγκόσμιο με το τοπικό. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια εξέλιξη στο ζήτημα. Μπορείτε να μου πείτε κατά πόσο η τοπική διάσταση μπορεί να παίξει μεγαλύτερο ρόλο. Σήμερα το διεθνές εμπόριο ενισχύεται, αφήνει όλο και περισσότερο χώρο στους, ε, σε όσους έχουν παρουσία σε πολλές αγορές. Ε, η, η, ε, η ψηφιακή διάσταση δίνει περισσότερες ευκαιρίες σήμερα, μπορεί κανείς να επεκτείνει τη δραστηριότητά του, αλλά τι θα κάνουν λιγότερο ανεπτυγμένες ή περισσότερο απομονωμένες περιοχές κατά την άποψή σας για να αναπτύξουν την επιχειρηματικότητα πράγματα θετικά για το εμπόριο δηλαδή, αλλά κάποιοι ακόμα δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα δίκτυα για να έχουν διεθνή παρουσία. Υπάρχουν δυνατότητες κατά την άποψή σας σε τοπικό επίπεδο. Πώς βλέπετε εσείς την κατάσταση που μεταβάλλεται ταχαίω σήμερα. Είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση σήμερα και εξελίσσεται διαρκώς. Ένα άλλο ζήτημα που μας απασχολεί αδιάκοπα είναι οι ευρωπαϊκές αξίες και η σχέση μεταξύ των δικών μα αξιών και των εμπορικών συμφωνιών. Έχουμε το παράδειγμα τη εμπορική συμφωνία με το Βιετνάμ. Εμεί προφανώ ε, ελπίζουμε η συμφωνία αυτή με το Βιετνάμ να μα δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στο Βιετνάμ. Ορισμένοι λένε ότι εξαιτία αυτών των ζητημάτων δεν έπρεπε να έχει συναυθεί εμπορική συμφωνία με το Βιετνάμ. Εσείς τι πιστεύετε. Ε, αυτοί οι κακοί μαθητές ε, ε, πρέπει να ε, πέφτουν θύματα αυτών των συμφωνιών. Πρέπει να ε, κάνουμε συμφωνίε με αυτούς τους κακού μαθητέ ή να του απομακρύνουμε. Ευχαριστώ. Κύριος Χέλμουτ Σούλτ. Ναι, ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε για αυτή την συζήτηση και ήθελα να σας ρωτήσω Τι σημαίνει σε εποχές ταραγμένες ε, αυτός ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου σήμερα, τι ρόλο μπορεί να παίξει. Παρότι ε, την προσοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Επιτρόπου ε, και του ανταγωνισμού με τις, Αμερι... Ε, με τις ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει την στρατηγική America First. Επιβάλλει τα δικά του κριτήρια για τα οικονομικά ζητήματα. Θα πρέπει λοιπόν να μας προβληματίσει η κατάσταση αυτή. Πώς θα διαμορφωθούν οι γραμμές παραγωγής, ε, οι υπηρεσίες, τα αγαθά που ανταλλάσσουμε με άλλες χώρες. Πώς θα τα καθορίσουμε όλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανάγκη, τις ανάγκες των ανθρώπων, ώστε να έχουμε μια οικονομία βασισμένη στις ανάγκες και αυτό να λαμβάνεται υπόψη στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και σε σχέση με τις κυκλικές οικονομίες. Να ξαναδούμε το γιατί εισάγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μήλα από την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία. Να δούμε γιατί ενθαρρύνουμε ορισμένους τρόπους κατανάλωσης. Αυτό που ήθελα να συζητήσουμε μαζί σας είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς σκέφτεται να αναδιοργανώσει τον τρόπο παραγωγής, κατανάλωσης και οργάνωσης του τρόπου ζωής μας λαμβανομένων υπόψεων των αναγκών αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, της πράσινης συμφωνίας κτλ. Αυτά πιστεύω διακυβεύονται διότι διαφορετικά θα συναγωνιζόμαστε να είμαστε ταχύτεροι, να πηγαίνουμε ψηλότερα, αλλά αυτό δεν είναι λύση. Αν πάτε να δείτε την Αυστραλία, βλέπετε τι έγινε εκεί. Εάν δεν δοθεί η ευκαιρία να οργανωθούμε κάπως και να ανταλλάξουμε απόψεις για το πώς θέλουμε να ζούμε και να ενσωματώσουμε αυτό στο εμπόριο και στην ανταλλαγή ε, αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ μας, δεν θα τα καταφέρουμε. Αυτό είναι κρίσιμο. Ε, ε, τώρα που ξεκινάει η δική σας θητεία, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια νέα στρατηγική διεθνούς εμπορίου. Εσείς ως Επιτροπή να την αναπτύξετε για να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανάγκες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Έχουμε μια ερώτηση από τον Μπεντ Λάγκε. Ε, κύριε Κότ. Αν κρατούσα μια... Αν σκεφτώ την απόσταση μεταξύ Αργεντινής και της χώρας μου. Και βλέπω να φεύγουν οι επενδύσεις ε, και βλέπω την παγκόσμια αλυσίδα αξιών να μην φέρνει ε, δουλειές στη χώρα μου. Και μετά ε, να έρχεται κάποιος και να μου λέει σας επιβάλλω και δασμούς. Σας επιβάλλω να τρώτε το δικό μου βοδινό για να ξαναφέρω τις επενδύσεις στη χώρα μου και για να αποσυνδέσω την αλυσίδα αξίας. για να βοηθήσω τη χώρα μου εναντί των ανταγωνιστών μου. Αυτή δεν θα ήταν μια στρατηγική επιτυχής. What do because we're really Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε ακόμα πέντε ερωτήσεις από τους ε, βουλευτές. Ε, μπορείτε να είστε σύντομοι, παρακαλώ. Βλέπω ότι έχουμε κάποια ε, κοινή θεματολογία θα μας δοθούν τελικές απαντήσεις βάσει αυτών των γενικών θεματολογιών, των γενικών θεμάτων που αναφέρθηκαν. Έχουμε την κυρία Ροντρίγκη Πινιέρο. Who που ήθελε να κάνει μια ερώτηση. <laughs> Muchas ευχαριστώ πολύ. Και ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα να φτάσω και ότι δεν μπόρεσα να ακούσω όλες τις παρεμβάσεις των εισηγητών. Σχέσεις Ευρωπαϊκή Ένωση, είπα. Όλοι θέλουμε να είναι αγαστές μέσα σε λογικά πλαίσια. Και για μας είναι λογικά πλαίσιο και ότι μπορεί να επιτευχθεί δηλαδή μία συμφωνία με σεβασμό στις αρχές που ε, στηρίζουμε μεταξύ αυτών και των, της, ε, της συμφωνίας του Παρισιού. Ήδη ο Ντόναλτ Τραμπ την έχει σχίσει τη συμφωνία αυτή. Εμείς πώς μπορούμε λοιπόν να διατηρήσουμε μια ισορροπία όταν λέμε ότι εμείς πρέπει να στηρίξουμε τις αρχές της, του Παρισιού ενώ ο Ντόναλτ Τραμπ ε, τις απορρίπτει παντελώς. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε σε άλλους, ας πούμε όπως η Βραζιλία, ε, που δεν μας ε, δίνουν κάποια αξιοπιστία εφόσον ε, δεν μπορούμε να στηρίξουμε τις αρχές αυτές. Δεύτερο ερώτημα, Κίνα. Εγώ είμαι υπέρ του να διατηρήσουμε μια λογική σχέση που να επιτρέπει την ε, ε, αντιστήχηση μεταξύ των δικών μας επιθυμιών και αυτών της Κίνας. Όμως υπάρχει ένα μεγάλο κεφόλιο, βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, θα ήταν δυνατόν να υπάρξει συνοχή σε σχέση με τα όσα εμείς λέμε στην εμπορική μας πολιτική. Και έπειτα, σχέση με αυτά που έλεγε η συνάδελφος Τσάμ, όσον αφορά την ενημέρωση των εμπορικών συμφωνιών, θα ήταν δυνατόν, λαμβάνοντα υπόψη ότι έχουμε κάνει βήματα μπροστά σε μια εμπορική πολιτική πιο φιλόδοξη, που συγκεντρώνει όχι μόνο τι είναι το ίδιο το εμπόριο, αλλά όλα τα μέσα της εμπορικής πολιτικής, ώστε να υπάρξει μια ενημέρωση με όχι τόσο περίπλοκο μέσο όπως ας πούμε η αναθεώρηση μιας εμπορικής συμφωνίας αλλά τουλάχιστον να δεσμευτούμε με όλες τις χώρες με τις οποίες έχουμε ήδη υπογράψει συμφωνίες να κάνουμε τη συμφωνία ότι θα στηρίξουμε η Συμφωνία του Παρισιού και να ξεκινήσουμε και με την αρχή ότι η προοπτική του φίλου θα λαμβάνεται υπόψη και στις εμπορικές συμφωνίες, ας πούμε, και για τη Χιλή, το εμπόριο, η Συμφωνία Εμπορίου με τη Χιλή, να, να είναι σαφές ότι το εμπόριο είναι για όλους. Μάλιστα. Ε, ωραία. Ο κύριος Ζουβά. Όχι, πρώτα, συγγνώμη, ο κύριος Χορδικάνιας. Ναι, ευχαριστώ. Ναι, το όνομά μου είναι μπερδεμένο, είναι δύσκολο, μην ανησυχείτε, μην ανησυχείτε, κανείς δεν το λέει σωστά. Νομίζω πως ε, είναι πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ακούσαμε σήμερα εδώ, όμως επιτρέψατε μου να σας πω μια σκέψη μου πριν από την ερώτηση. Είμαστε σε μια φάση όπου τα αξιώματα με τα οποία έχουμε δουλέψει μέχρι στιγμής αμφισβητώνται. Το εμπόριο, ενώ είναι καλό, λέγαμε παλιά, για πολλούς φαίνεται όμως πως όχι πια. Αμφισβητείτε το εμπόριο. Όχι από τους ε, παλιούς ε, και τους ε, ανέκαθεν εχθρούς του εμπορίου, αλλά και από αυτούς οι οποίοι είναι υπέρ του καμουφλαρισμένου προστατευτισμού και προσπαθούν να μην συζητήσουν για τις δυσκολίες, τις βελτιώσεις του ίδιου του εμπορίου των μέσων με βάση δεδομένα, αλλά με βάση τις ε, ζημιές και την ιδεολογία. Αυτό είναι θεμητό, όμως μέσα στη συζήτηση μπαίνει και ένα στοιχείο το οποίο δύσκολα μπορούμε να ξεπεράσουμε, τουλάχιστον με βάση τα όσα ε, διαβάζω. Και σας έλεγα, δεν μπορούμε να το δούμε βραχυπρόθεσμα το θέμα, θα πρέπει να σκεφτούμε διορατικά για στο εμπόριο, το πώς θα μπορέσει όλος να μας ωφελήσει, όχι μόνο για να προχωρήσουμε και να αυξήσουμε την ευημερία, αλλά να αποτελέσει ένα μέσο, ένα μέσο, όχι το μοναδικό, που θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε κάποιους στόχους περιβαλλοντικούς, αναπτυξιακούς κτλ. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα, ότι δηλαδή τα πολιτικά ωφέλη τα παίρνει κανείς βραχυπρόθεσμα. δεν, γίνονται, δεν επενδύονται μακροπρόθεσμα. Άρα λοιπόν, σε σχέση με μια συζήτηση για το τι είδου εμπόριο θέλουμε να αναπτύξουμε σε Ευρωπαϊκή Ένωση, που μάλλον θα πρέπει να το αναπτύξουμε υπό το φω τη Νέα Συμφωνία, του Πράσινου Συμφώνου, βλέπουμε πω μέσα στο ίδιο το Κοινοβούλιο γίνεται συζήτηση όπου όταν αμφισβητείται η εφαρμογή του Πράσινου Συμφώνου και η επιρροή αυτή στην εμπορική συμφωνία, στι εμπορικέ συμφωνίε και γενικότερα στο εμπορικό ε, παγκόσμιο μοντέλο. Όχι, ας πούμε, βλέπουμε πώς θα επηρεάσει το πράσινο σύμφωνο τη Μερκοσούρ. Γιατί, γιατί περάσαμε το TTP, κακήν κακό, τη ΣΕΤΑ κακήν κακός και τώρα είμαστε στη Συμφωνία Μερκοσούρ. Είναι λοιπόν απαραίτητο να δούμε πώς θα ε, εξυγχρονίσουμε το μοντέλο του εμπορίου μας, για ποιο λόγο θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε, τι κόστο και τι όφελο θα μα αποφέρει για όλου. Γιατί υπάρχουν ε, και μέρη του κόσμου που μπορεί να πούνε «Α, εμείς δεν θέλουμε, πάμε με την Κίνα να συνεργαστούμε» π.χ. Αυτό θα πρέπει να το δεχτούμε, ότι ορισμένε από τι απαιτήσει μα μέσα σε αυτέ τι εμπορικέ συμφωνίε μπορεί να σημάνουν προβλήματα. Εγώ δέχομαι πω είναι απαραίτητο, γιατί το δικό μα μοντέλο ε, εμπορίου θα πρέπει όλα αυτά να τα ε, περιλαμβάνει. Ε, πρέπει να είμαστε υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης, ε, της μη επιρροής, της μη αρνητικής επιρροής στην ε, οικολογία και στο περιβάλλον, αλλά με βάση συγκεκριμένα δέδομα. Και για να τελειώνω, είναι περίπλοκο το θέμα να συζητάμε σε εθνικό επίπεδο για μια συμφωνία, όταν οι περισσότεροι που το συζητούν, τη συζητούν τη συμφωνία αυτή δεν έχουν καν διαβάσει. Πώς μπορούμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Big λίγο μεγάλο αυτό το ερώτημα. Κύριε Ζουρδά, ευχαριστώ. Να σας διαβεβαιώσω ότι η δική μου ερώτηση θα είναι πολύ πιο σύντομη. Διαπιστώνω κάτι πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το πάνελ και έχει σχέση το ερώτημά μου με τις πρακτικές των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην επαγγελματική μου πρακτική έχω διαπιστώσει την προσπάθεια των ΗΠΑ να επιβάλλουν έξω εδαφικά την ομοθετησία τους και την περιφρόνησή τους για το διεθνές δίκαιο. Έχω ζήσει εγώ την, τον εκφοβισμό ουσιαστικά προσπαθώντας από τις Ηνωμένε Πολιτείες ε, ή, από, ε, που προσπαθούν μάλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες ή κάποιες επιχειρήσεις τους να ασκήσουν για να αποκτήσουν οικονομικά ωφέλη. Το ερώτημα λοιπόν είναι, αφού μιλούμε ε, για την σημασία της πολυμερούς διαπραγμάτευσης, αρκεί αυτό και αν ναι, πώς θα βρούμε συμμάχους για να αλλάξουν τα πράγματα και ουσιαστικά για να περιορίσουμε αυτήν την μονομερή προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών και πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε μια συμμαχία η οποία να αλλάξει το συσχετισμό δυνάμεων υπέρ μας ή μήπως είμαστε καταδικασμένοι απλώς να συνεχίζουμε με ομορφά λόγια αλλά στην πραγματικότητα να υποκείμεθα σε αυτό τον ε, αμερικανικό, την αμερικανική επιβολή. Έχω δύο ερωτήσει, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Είναι γνωστό ότι η τελευταία γενιά συμφωνιών ελευθέρω εμπορίου που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτε χώρε. συμπεριλαμβάνουν και πολλά άλλα πράγματα εκτό από ζητήματα εμπορίου. Και δεν μιλώ μόνο για το TSD, αλλά επίση και για τι συμφωνίε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τι συμβάσει του ε, Διεθνούς Οργανισμού Εργασία κτλ. Επομένω, ήδη απαιτούμε πολλά από του εταίρου μα ενώ υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες απαιτούν πολύ λιγότερα. Όλοι στο πάνελ ουσιαστικά αναφέρατε ότι θα πρέπει να αγωνιστούμε έτσι ώστε σε παγκόσμιο επίπεδο να υπάρχει ισότιμο ανταγωνισμός, γιατί αυτό θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις μας. Όμως η πραγματικότητα είναι λίγο πιο περιπλόκη. Και θα ήθελα να μου πείτε τι πιστεύετε εδώ. Δεν πιστεύετε ότι υπάρχει μια κάποια αντίφαση. Μήπως η νοοτροπία που έχουμε υιοθετήσει στα ζητήματα των εμπορικών συμφωνιών δεν βοηθάει την ανταγωνιστικότητά μας, μήπως την πραγματικότητα βλάπτει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Πρόσφατα διάβασα ένα άρθρο του Bloomberg, στο οποίο αναφέρεται ότι περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια θα χάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτία της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, η οποία μόλις συνήφθη την πρώτη φάση της συμφωνίας. Και ότι λέει το άρθρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει κατά πόσον αυτή η συμφωνία είναι συμβατή με τους κανόνες του ΠΟΕ. Συμφωνείτε με αυτή την αξιολόγηση η οποία για την ακρίβεια την δημοσιεύει το Bloomberg αλλά έχει προέλθει από ένα γερμανικό Ινστιτούτο Μελετών. Συμφωνείτε εσείς με αυτή την εκτίμηση των πραγμάτων. Τελευταία ερώτηση, κύριε Κόνσοπλ. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετική ημέρα για το διεθνέ εμπόριο σήμερα. Γιατί, γιατί σήμερα το πρωί εγκρίναμε τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με το Βιετνάμ και τώρα το απόγευμα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αυτές τις εξαιρετικές παρουσιάσεις των συμμετεχόντων στο πάνελ μας. Και αυτό είναι τον ε, εναρκτήριο λόγο της κυρίας ε, Βάινερ που ήταν εμπνευστικός. Είναι πολύ σημαντικό να εργάζεται κανείς στο ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί προσπαθούμε μεταξύ μας να συνεργαστούμε για να επιλύσουμε παγκόσμια προβλήματα. Και βέβαια, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε διεθνώς είναι η μείωση της εξάρτησής μας από τα όρεκτα καύσιμα και η μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Άλλη μία πρόκληση είναι να πάψουν οι ε, Ενισχύσει ε, προς συγκεκριμένου κλάδους ε, της βιομηχανίας ή της οικονομίας. Ε, και θα πρέπει να δούμε πού συμπλέκονται αυτά τα δύο ζητήματα. Οι κρατικές ενισχύσεις για την χρήση ορυκτών καυσίμων, που είναι ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα, αλλά πολύ σημαντικό για την κλιματική αλλαγή. Θα μπορούσατε λοιπόν ε, ακόμα και τώρα αργά το απόγευμα να μου πείτε, από τις δικές σας γνώσεις και εξειδικευμένη εμπειρία, πώς μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα από, ε, από την οπτική γωνία του, ε, της εμπορικής πολιτικής. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Σας ευχαριστούμε. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας και θα αξιοποιήσω και την ιδιότητά μου συντονίστρια Πολλά από αυτά τα ζητήματα που τέθησαν έχουν σχέση με τον ΠΟΕ και την ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Θα σας πρότεινα όμως όλα αυτά τα ερωτήματα να μην τα συζητήσουμε τώρα, να πάνε για το επόμενο πάνελ που είναι ακριβώς για το θέμα αυτό. Θα ζητήσω λοιπόν από τους ομιλητές μας να απαντήσουν. Ένα θέμα που είδα να έρχεται και να ξανάρχεται είναι το εξής. Τι μπορούμε να πετύχουμε στην πραγματικότητα ε, πώς μπορούμε να ελέγξουμε τις, με τις Ηνωμένες μπορούμε να ελέγξουμε τις Ηνωμένε Πολιτείε. Πώς μπορούμε να ε, ελέγξουμε δύσκολους εταίρους. Τι μπορεί να επιτευχθεί τη χρονιά αυτή. Ένα δεύτερο μεγάλο ερώτημα είχε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο επικοινων... δημοσιοποιούμε την εμπορική μας πολιτική, πώς επικοινωνούμε με τις διάφορες Κοινωνικέ ομάδε, διαφορε περιφέρειες οι οποίες μπορεί να αισθάνονται ότι υπονομεύονται ή τις αγνοούμε. Και αυτό συνδέεται με όλη τη συζήτηση για την σχέση της εμπορικής πολιτικής με την κυριαρχία. Τσούλια, μήπως θέλετε να ξεκινήσετε εσεί. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και δύσκολες. Για τις ροές δεδομένων πιστεύω αυτό που έχουμε δει Έχουμε δει σε 160 χώρες περίπου 45 δεν έχουν τίποτα. Πρέπει να επιλέξουν. Υπάρχουν πολλές χώρες που κυρίως ανησυχούν για θέματα ιδιωτικού απορρίτου και άλλες έχουν πολλούς περιορισμούς είτε βασισμένους σε κάποια ιδιαίτερη άποψη για τη βιομηχανική πολιτική ή για την ασφάλεια. Θεωρούν ότι αν κρατήσουν τα δεδομένα δικά τους τότε θα αναπτυχθούν βιομηχανικά. Όταν λέτε λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι μικρότερο, πρέπει να γίνει μικρότερο του ψηφιακού, ναι, υπάρχουν φιλοσοφικές, ιδεολογικές διαφορές ε, για το ιδιωτικό ε, απόρριτο και για τον προστατευτισμό. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να καταλάβουμε πώς ε, μεταβιβάζουν δεδομένα οι επιχειρήσεις, ποιες διατάξεις απορρίτου εφαρμόζονται και να προσπαθήσουμε τι ομοιότητε υπάρχουν. Αν δούμε του κανονισμού σε εθνικό επίπεδο σε πολλέ χώρε υπάρχουν περισσότερε ομοιότητε από ό,τι θα πίστευε κανεί. Οπότε είναι δύσκολο το έργο αυτό, αλλά πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να αποκομίσουμε τα ωφέλη. Να αφήσουμε δηλαδή την ευρεία ιδεολογική περιγραφή και να προσπαθήσουμε να βρούμε τι συμβαίνει πραγματικά, ούτω ώστε κάποια από τα ωφέλη, ειδικότερα για τι μικρέ επιχειρήσει και για τι γυναίκε, να γίνουν πραγματικότητα. Διότι τίποτα δεν θα επιτευχθεί αν δεν μπορεί κανείς να διαβιβάσει δεδομένα. Τώρα για τις περιφερειακές, για τις απόμακρες περιοχές. Ξέρουμε πολλές περισσότερες επιχειρήσεις ε, που εμπλέκονται στο διεθνές εμπόριο, παρέχοντας ε, ε, προϊόντα σε μικρές επιχειρήσεις, τοπικές επιχειρήσεις που εξάγουν. Οπότε υπάρχει και αυτό και είναι μεγάλο κομμάτι του διεθνούς εμπορίου. Κάτι άλλο. για την Πράσινη Συμφωνία είναι πολύ σημαντικό και θα συζητηθεί πολύ. Υπάρχουν πολλά περιθώρια για να κερδίσουν όλοι από τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες στην κυκλική οικονομία. Θα γίνει και μια ενδιαφέρουσα και δύσκολη συζήτηση όμως για το τι, ποια είναι η χρηστή επιχορήγηση και ποια πράσινη επιχορήγηση θα είναι καλή. Κανείς δεν επιχορήγει λέγοντας θα δώσω ένα καρό λεφτά σε συγκεκριμένα συμφέροντα. Όλοι λένε ότι θέλω να εξυπηρετώ κάποιο σκοπό. Οπότε α κάνετε, διαχωρίσετε το τι, ας διαχωρίσουμε το τι λειτουργεί και το τι είναι σημαντικό. Ξέρουμε ότι κάποιε επιχορηγήσει δεν είναι καλέ. Οι επιχορηγήσει στα ορεικτά καύσιμα δεν είναι καλέ, είναι επιβλαβεί. Έχουμε επιχορηγήσει στην Αλία που συμβάλλουν ε, στην υπεραλίευση. Οπότε συμφωνώ μαζί σα. Θα είναι σημαντική αυτή η συζήτηση, αλλά είναι και συζήτηση που πρέπει να γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί κάποιε επιλογέ επηρεάζουν το εύρο επιλογών που έχουν και οι χώρε. Και πιστεύω ότι αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ στενά και πολύ σοβαρά το πώ θα μπορέσουμε να μειώσουμε τι καθαρέ παγκόσμιε εκπομπέ. Γιατί ενίοτε δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζουμε. μένα μου αρέσουν οι ντομάτε, α πούμε. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα. Ε, πώ θα τι φάει κανεί στην Νορβηγία στα μέσα του χειμώνα. Ναι, το, το, και αυτές παράγονται εκεί, σε θερμοκήπια, δεν είναι περιβαλλοντικά φιλικές. Τώρα για τη δημόσια υποστήριξη, ναι, πολύ περισσότερο κόσμος τώρα ε, βλέπει πιο θετικά το εμπόριο γιατί είναι πολυμερές. Αλλά και ο οικονομικός εθνικισμός είναι κάτι που αποτελεί πλέον πραγματικότητα. Δύο πράγματα πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε εύκολα τις εναλλακτικέ ειδήσει ή τι προκαταλήψει, αλλά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάποιους ανθρώπους, που αντιμετωπίζουν κάποιοι άνθρωποι και οδηγούνται σε οικονομικό εθνικισμό. Θα κλείσω με το πώς θα καταφέρουμε την πολυμερή προσέγγιση Έχω διάφορες ιδέες. Κάποια από τα ζητήματα προσπάθησα να θίξω εγώ είναι αυτά που προσπαθούμε να υπογραμμίσουμε σε όσου ε, μιλούν για πολυμερή προσέγγιση. Αν δούμε τη συμφωνία μεταξύ ΙΠΑ και Κίνα, αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι δεν ασχολήθηκε κανεί με τι επιχορηγήσει, Ενώ είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Οπότε πρώτον ας ε, μιλήσουμε καθαρά για κάποια ζητήματα. Α μην κάνουμε τα στραβά μάτια. Μετά οι σύμμαχοι. Υπάρχει μια συμμαχία, πιστεύω, ένα συνασπισμό αναπτυγμένων περιοχών, ε, χωρών. αλλά αυτοί που θα υποφέρουν από έναν πόλεμο επιχορηγήσεων, από τις μεγάλες ενδεχομένως δυνάμεις, ε, ε, θα είναι οι οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες και οι ανεπτυσσόμενες χώρες. Έχουμε, ξέρετε, υπάρχει πολυμερής προσέγγιση και στην Αμερική, αλλά αυτοί δεν έχουν την εξουσία σήμερα. Υπάρχουν μεταρρυθμιστές στην Κίνα, ε, αλλά δεν έχουν δύναμη αυτή τη στιγμή. Πώς θα επικοινωνήσουμε μαζί τους. Υπάρχουν και πολλά εργαλεία. Η Airbus και Boeing ήταν μια, ένα πολύ καλό παράδειγμα Οι νομικοί τα παράτησαν, μετά από τόσα χρόνια διαπραγμάτευσης πήγαν στα γιο τους και τώρα είμαστε ξανά στη διαπραγμάτευση που είναι χαρακτηριστικό της πολυμερούς προσέγγισης. Οπότε διαφάνεια στις συμφωνίες. Πρέπει να προσέξουμε να μην πηγαίνουμε προς τα πίσω. Όλη αυτή η πολυμερή συνεργασία που έχουμε απλά Ξέρετε, όταν συμπεριφέρεται κανείς κακά, προκαλεί κακές συμπεριφορές. Οπότε, να παραθέσω αυτά που είπε ένας παλιότερος Αμερικανός πρόεδρος. Κάνω ό,τι μπορείς, όπου βρίσκεσαι με αυτά που έχεις. Ευχαριστούμε πολύ, ρεαλιστικό συμπέρασμα. Πιτ, ε, ακούσα, υπήρχαν ερωτήσεις για σας. Ευχαριστώ πολύ ε, και την πρόεδρο. Και ο πρόεδρος έκανε πολλές ερωτήσεις. Ε. Φυσικά γνωρίζουμε και εγώ δεν υποστήριζω την επιστροφή σε οικονομία διαβίωσης. Οι παγκόσμιες αλυσίδες ε, προμηθειών είναι πραγματικότητα. Η οικονομία μας είναι παγκοσμιοποιημένη. Η παγκόσμια οικονομία. Καμία χώρα δεν μπορεί να ε, απομονωθεί χωρίς να υποστεί τεράστια βλάβη. Επίσης, ε, το κύριο ερώτημα είναι ο κόσμος ακόμα υποστηρίζει το εμπόριο. Είναι ισχυρότεροι αυτοί που αντιτίθεται στο εμπόριο από αυτού που το υποστηρίζουν. Δεν ξέρω την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, αλλά αυτό μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι πρέπει να ξεχάσουμε την παλιά νοοτροπία που έλεγε ότι κάθε απελευθέρωση του εμπορίου είναι εξορισμού καλή και ότι οποιασδήποτε εταιρείε, ε, περιοχές, ε, οποιοδήποτε εργοδότες και εργαζόμενοι ε, που υφίστανται κακές συνέπειες του εμπορίου ε, υποφέρουν από αυτό λόγω προβλημάτων ανακατανομής που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε τοπικό επίπεδο. Πιστεύω ότι πρέπει να εξελίξουμε κάπως τον τρόπο σκέψης μας ε, και να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές, τα πραγματικά αποτελέσματα και σε θέματα ανακατανομής για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια εμπορική πολιτική που θα πείσει τον κόσμο ότι του συμφέρει. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα από τη δική μου περιοχή η διαιτησία για τις επενδύσεις ε, αμφισβητήθηκε πολύ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ως νομικός εγώ ε, πρέπει να σας πω ότι δικαίως το σύστημα αυτό χρήζει μεταρρύθμισης. Λειτουργεί περισσότερο προς όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων παρά άλλων ε, συμφερόντων που επίσης χρήζουν προστασίας. Οπότε πρέπει να εστιαστούμε πιστεύω στο γεγονός ότι οι διαφορετικές εμπορικές πολιτικές ε, έχουν διαφορετικά αποτελέσματα και έτσι η απελευθέρωση του εμπορίου δεν αφορά μόνο την αύξηση του ΑΕΠ και των εξαγωγών, αφορά και το τι γίνεται επί τόπου. Σχετίζεται με το ζήτημα της βιωσιμότητας και με το κατεπήγον ζήτημα του κλίματος. Κάποιες μορφές εμπορίου είναι πολύ καλές για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του κλίματος, αλλά άλλες μορφές εμπορίου δημιουργούν πρόβλημα. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Η Άννα Στέλιγκερ. Ε, κοιτάξτε, απάντησαν σε πολλέ ερωτήσει ήδη οι συναδέλφοι και συμφωνώ με τα όσα είπε η Τζούλια Νίλσεν για τα δεδομένα και την ελεύθερη ροή δεδομένων και την ψηφιοποίηση, για παράδειγμα. για το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο και για την άποψη για το εμπόριο. Αν δούμε τα τελευταία νούμερα της Eurostat, η υποστήριξη για το εμπόριο αυξάνεται στις περισσότερες χώρες. Στη δική μου χώρα ε, είναι στο 86%. Είναι η υψηλότερη υποστήριξη του παγκοσμίου εμπορίου που υπάρχει σε οποιαδήποτε χώρα. Στην Ιταλία είναι μεταξύ 35 και 40. Είναι λοιπόν πολύ κατακαιρματισμένη εικόνα στην Ευρώπη όσον αφορά την κοινή γνώμη για τα ωφέλη του εμπορίου. Πιστεύω ότι έχουμε τεμπελιάσει. Μιλάμε για διεθνές εμπόριο όταν ο ΠΟΕ έχει ένα, υποστή παράλυση στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο. Μιλάμε για τη λειτουργία του διεθνού εμπορίου, ενώ έχουμε παγκόσμιε διενέξει. Και μιλάμε για τα ωφέλη τη εσωτερική αγορά, ενώ ζούμε και τον Brexit ταυτόχρονα. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε πια να τεμπελιάζουμε, δεν έχουμε τέτοιο περιθώριο. Θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση για τα μακροχρόνια και τα βραχυχρόνια εκτίματα για να εξηγήσουμε τι είναι το εμπόριο, τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί. Τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις. Μπορούν να δεσμευτούν, να διευκολύνουν και να ασκήσουν πίεση. Θα πρέπει να διευκολύνουμε κάποια πράγματα τα οποία σχετίζονται με το επόμενο πάνελ που έχει να κάνει με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει να διευκολύνουμε την πράσινη καινοτομία, να άρουμε τα εμπόδια για την κυκλική οικονομία. Υπάρχουν εμπόδια για την ανακύκλωση υλικών, για παράδειγμα, για την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων αντικειμένων. Θα πρέπει να άρουμε αυτά τα εμπόδια και για το πράσινο εμπόριο, για την κυκλική οικονομία. Καθημερινά συναντάμε εταιρείε που μα λένε ότι έχουν καταπληκτικέ ιδέε ε, για το επιχειρηματικέ, ε, ε, φιλικέ προ το περιβάλλον, αλλά αντιμετωπίζουν εμπόδια. Θα πρέπει να τι βοηθήσουμε. Επίση, να ασκήσουμε πίεση για κάποιε διαπραγματεύσει. Έχουμε μία συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά που είναι εντάξει αυτή τη στιγμή, αλλά έχει τελματώσει. Χρειαζόμαστε τέτοιε διαπραγματεύσει και το ξέρουμε. Επίση, πρέπει να συμπεριλάβουμε τι υπηρεσίε ε, στη συμφωνία για τις, ε, τα περιβαλλοντικά αγαθά. Πόσο δύσκολο είναι. Επίση, θα πρέπει να δεσμευτούμε. Και εδώ θέλω να κάνω τον παραλληλισμό με τον ΠΟΕ. Ξέρουμε ότι ο σχετικό γύρο συζητήσεων έφερε αποτελέσματα. Ο λόγο ήταν ότι οι υπηρεσίε άσκησαν πίεση ε, στο Euroground και στον ΠΟΕ για να φέρει αποτελέσματα. Δεν βλέπω να γίνεται αυτή τη στιγμή ιδιαίτερη πίεση στο σημερινό ε, γύρο του ΠΟΕ. Πρέπει να είμαστε παρόντες, να ασκήσουμε πίεση και να άρουμε τα εμπόδια ε, για το πράσινο εμπόριο και να καταστήσουμε το εμπόριο ε, θέμα που να, μένει, να έχει νόημα στην ατζέντα της βιωσιμότητας. Κοιτάξτε την ατζέντα του 2030. Προφανώς το εμπόριο δεν είναι το μόνο εργαλείο, αλλά είναι ένα από τα εργαλεία χωρίς το οποίο δεν μπορούμε να βελτιώσουμε τον κόσμο μέχρι το 2030. Ευχαριστούμε πολύ, Σαμπίνε. Ένα λεπτό. Το λέω γιατί είμαι βέβαιο ότι θα επανέλθετε στην Επιτροπή μας και θα επανέλθετε συχνά, αλλά όχι άλλοι Οπότε... Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν έχω να πω πολλά. Συμφωνώ με τα περισσότερα που είπαν οι, προ... οι υπόλοιποι πανελίστες. Ε, ο Πίτερ Εκχάουτ είπε ότι έχουμε το πλεονέκτημα ότι είμαστε λογικοί και ότι δεν παίζουμε το λαϊκιστικό παιχνίδι. Ταυτόχρονα, ωστόσο, αυτό, ξέρετε, είναι τόσο ισχυρό όσο και αδύναμο σημείο. Είναι αδύναμο σημείο όταν συζητάμε δημοσίω. Ο μόνο τρόπο ε, που έχουμε στα χέρια μα είναι να παρουσιάσουμε τα γεγονότα και να κάνουμε μια συζήτηση βάσει πραγματικών στοιχείων. Αλλά σε ένα ιδεολογικά φορτισμένο περιβάλλον, το να ακουστεί κανεί μέσα σε τόσο σαματά είναι εξαιρετικά δύσκολο. Αυτό το έχετε ζήσει και εσεί ω βουλευτέ. Αυτό εξηγεί ενδεχομένω και την στρέβλωση στη δημόσια συζήτηση. Αφενός ε, έχουμε αύξηση των ανθρώπων που βλέπουν θετικά το εμπόριο, αλλά δεν κατεβαίνουν αυτοί στους δρόμους. Αυτοί που κατεβαίνουν στους δρόμους είναι πολύ πιο κινητοποιημένοι, αντίθετοι προς το εμπόριο. Και αυτό μας φέρνει σε μια κατάσταση όπου αρχίζουμε να μιλάμε τελικά μόνο για τα πλεονεκτήματα των πολιτικών μας τη στιγμή όπου υπάρχει κίνδυνο να τα χάσουμε. Και αυτό είναι το πρόβλημα που θα πρέπει να εξετάσουμε μαζί. Και εγώ δεν έχω απάντηση γι' αυτό. Είναι δύσκολη δουλειά. και δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, πρέπει να προκαταβολικά να αναφέρουμε ποιο είναι το κόστος και τα ωφέλη του εμπορίου, να εξετάζουμε φυσικά την κατανομή όλων αυτών και να ξέρουμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Αλλά η εμπορική πολιτική επίσης θεωρείται υπεύθυνη για όλα τα προβλήματα που δημιουργεί η ψηφιοποίηση σε τεχνολογικό επίπεδο. Και η απάντηση εδώ δεν μπορεί να δοθεί μόνο από την εμπορική πολιτική. Το δύσκολο είναι η ολοκλήρωση των πολιτικών. Και το τελευταίο που έχω να πω για όλα αυτά, όταν μιλάμε για συνοχή τη πολιτική, ε, όταν συζητάμε για το πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τι ε, περιβαλλοντικά επιζήμιε επενδύσει, ε, επιχορηγήσεις, συγγνώμη. Ε, εδώ δείτε μέσα στο κοινοβούλιο πρόσφατα ψήφισε να ενισχυθούν οι επιδοτήσεις για την αλληλεία, ενώ εμείς στη Γενέβη προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τι περιορίσουμε αυτέ τι επιχορηγήσει. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το δούμε πώς θα το κάνουμε όλοι μαζί. Ευχαριστούμε πολύ. Εξαιρετική εισαγωγή για το επόμενο πάνελ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε και το γεγονός ότι είχαμε τόσους βουλευτές που έθεσαν ε, κέρια ερωτήσεις σημαίνει πως έχουμε πολλά ακόμα να συζητήσουμε και να κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Okay, so uh, in the of time we are to the next panel. Μάλιστα, πολύ ωραία. Περνάμε στο επόμενο πάνελ. Ε, ε, έχουμε τώρα μια συζήτηση για την πτυχή της βιωσιμότητας σε σχέση με την εμπορική πολιτική. Από την προηγούμενη ε, συνεδρία είδαμε ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε την ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική και τους στόχου βιώσιμη ανάπτυξη. Αν εγκαταλείπετε την αίθουσα, παρακαλώ εγκαταλείψτε την ισιοπυρό. Σας ευχαριστώ πολύ. Το καλό και το κακό ταυτόχρονα είναι ότι έχουμε μόνο τρεις ομιλητές. Έχουμε έναν καλό ομιλητή που δεν μπόρεσε να είναι παρόν, ε, ε, ομιλήτρια, την κυρία Εβίτα Αλλά αυτό σημαίνει πως θα έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε τα όσα θα συζητήσουμε. Ε, έχετε υπόψη ότι στις 6 ακριβώς ε, θα πρέπει να τελειώσουμε και να εγκαταλείψουμε την αίθουσα. Έχουμε λοιπόν ε, την Ιζαμπέλ Ντουράν, αναπληρωματική γενική γραμματέα της UNCTAD, στον ΟΙΕ έχουμε τον Καλ Μπράουνερ που είναι αναπληρωτής ε, Γενικός Διευθυντής του ΠΟΕ και μπορεί να απαντήσει και όλα σε ορισμένα από τα ερωτήματα που ήδη τέθηκαν νωρίτερα. Και έχουμε και τον Μάρκ Μάις που είναι υπεύθυνο συμπορικής πολιτικής στην Βελγική ΜΚΟ 11-11-11 να μας πείτε δύο λόγια και για το τι κάνετε. Βασικά λοιπόν έχουμε να συζητήσουμε την εμπορική πολιτική και πώς μπορεί να συμβάλλει στην ε, ατζέντα των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Ιζαμπέλ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω γαλλικά. Le commerce va servir euh, les objectifs du développement durable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 Ε, αλλάξει η κατάσταση και το εμπόριο θα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα. Αυτά όλα λοιπόν είναι προκλήσεις. Προκλήσεις ε, στις κλιματικές, ε, είναι κλιματική αλλαγή στις οποίες θα πρέπει να προσαρμοστεί και το εμπόριο. Θα πρέπει να οργανωθούμε για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε. Τέλος, πολυμερή συνεργασία. Υπόθηκε και στην προηγούμενη συνεδρίαση ότι δηλαδή ορισμένες συμμαχίε που βγαίνουν από την πεπατημένη, που δεν πολλώνουν τα πράγματα ανάμεσα στους καλούς και τους κακούς, την κλασική εικόνα και την εικόνα που εργάζεται με συγκεκριμένες συμφωνίες, θα μπορούσε να βοηθήσει στο να σωθεί η πολυμερή συνεργασία ή, εν πάση να δημιουργηθούν διαφορετικέ συμμαχίε για δεδομένα θέματα, όχι απαραίτητα για όλα, γιατί υπάρχουν ε, πράγματα τα οποία διχάζουν. Αλλά, ας πούμε, στο ψηφιακό τομέα και στις κλιματικές αλλαγές είναι δύο πράγματα, δύο θέματα όπου μπορούμε να βγούμε συμμαχίες ώστε να ε, δώσουμε περισσότερο χαρακτήρα στην πολυμερή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ευχαριστώ και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε, είδη, κάθε θέμα που εμπίπτει στις δικές μας αρμοδιότητες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την αισιόδοξη διάσταση και δημιουργική προσέγγιση που είχε η παρουσίασή σας. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Καρλ Μπάουνα. Τι μπορεί να κάνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου για του βιώσιμους στόχους, για βιώσιμης ανάπτυξης, τι κάνει ήδη και τι μπορεί να βελτιώσει. Σα ευχαριστώ πρώτα απ' όλα να σα ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Πάντοτε είναι, είμαι ευτυχή όταν επισκέπτομαι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε 17 στόχου βιώσιμη ανάπτυξη από εκείνου που έχει καθιερώσει ο ΙΕ που μπορούν να του υποστηρίξουμε μέσω του διεθνού εμπορίου. Εγώ θα αναφερθώ στον 14-6 που αναφέρεται στις, στην υποστήριξη της αλληλεία έχει δοθεί στον ΠΟΕ η αρμοδιότητα για την διαπραγμάτευση των ε, ε, επιδοτήσεων της Αλίας και για άλλη μια φορά οι υπουργοί στη σχετική υπουργική διάσκεψη συμφώνησαν ότι μέχρι το 2020 θα έχουν καταργηθεί ορισμένες μορφές επιδότησης της Αλίας οι οποίες οδηγούν σε υπεραλίευση και να σταματήσουν οι επιδοτήσεις εκείνες οι οποίες οδηγούν σε παράνομη αδήλωτη ε, ε, ανεξέλεγκτη αλεία. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει ο ΠΟΕ σε τέτοιες διαπραγματεύσεις και είμαι ιδιαίτερος ευτυχής που είμαι αναπληρωτής διευθυντής των ΠΟΕ και προέρχομαι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ο ΠΟΕ είναι μία από τις λίγες ε, διεθνείς οργανώσεις που συνεχίζει να προσπαθεί να προωθήσει το κοινό, τα κοινά αγαθά παγκοσμίω, όπως για παράδειγμα τα αλλιευτικά αποθεύματα μας θάλασσες και τους ωκεανού μα. Έχει λοιπόν την εξειδικευμένη γνώση για τα ζητήματα των επιδοτήσεων ο ΠΟΕ. Θα έλεγα ότι ο στόχος 14-6 δεν είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος, μιλούμε μόνο για υπεραλίευση, μιλούμε για την κατάρκηση των επιδοτήσεων μόνο που, εκείνων που οδηγούν σε ε, αδήλωτη και παράνομη αλία. Όμως θα ήθελα να συνδέσω την παρουσίασή μου με αυτά που έλεγε και η κυρία Βάιναντ προηγουμένως για να σας παραπέμψω στο, σε μια άλλη δέσμευση στο 14.6 λέγεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση να μην υιοθετηθούν, να μην ε, ε, δημιουργηθούν ε, τέτοιες ενισχύσεις είχε ένα πρόγραμμα η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντικατάσταση των παλαιών σκαφών του στόλου. Ε, το προηγούμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η προηγούμενη θητεία, εν πάση περιπτώσει, επαναβεβαίωσε τη, συνε... τη συνέχιση του προγράμματος. Εγώ δεν θέλω να αξιολογήσω το πρόγραμμα αυτό, όμως το μόνο που θα ήθελα να κάνω εδώ σήμερα είναι να εφιστήσω την προσοχή σα στο γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται στο διεθνές επίπεδο ως υπόδειγμα, ως μία έλογη δύναμη, ως εκείνη η δύναμη την οποία θα πρέπει να ακολουθούν όλες οι χώρες που θέλουν να κάνουν το ηθικά σωστό. Επομένως οτιδήποτε και αν αποφασίζεται θα πρέπει να δημοσιοποιείται με τέτοιον τρόπο που να μην δίνει μια λανθασμένη ε, αντίληψη, λανθασμένο μήνυμα στις διαπραγματεύσεις στη Γενέβη. Και αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο γιατί φανταστείτε εκείνους τους εκπροσώπους των κρατών που ε, διαπραγματεύονται για ζητήματα επιδοτήσεων στην Αλία στη Γενέβη, αυτοί μπορεί να καταλήγουν στις δικές τους ε, θέσεις με βάση ε, μια υπεραπλουστευμένης ορισμένης περιπτώσεις ανάλυση της πραγματικότητας. Γνωρίζουμε ότι μια σωστή αντίληψη της πραγματικότητας πρέπει να βασίζεται σε πλήρη στοιχεία και αυτό δημιουργεί πάντοτε προβλήματα και δυσκολίες. Δυστυχώς, η νοτροπία των καιρών μας δεν προάγει τη συνεργασία. Και αυτό ίσως φαίνεται και στο γεγονός ότι χρειάστηκαν πέντε μήνες να ε, διαπραγματεύσεων για να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη του ΠΟΕ ε, στον ορισμό ενός νέου Προέδρου για την Επιτροπή. Ε, και το οποίο συνέβη μόνο όταν απεμπόλησε ένα άλλο αξίωμα στη χώρα του άνθρωπος αυτός, το οποίο σημαίνει και μας δείχνει πόσο σημαντική είναι η προσπάθεια, θα είναι η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καθοδηγήσει τις διαπραγματεύσεις αυτές προς μια αίσια έκφαση. Ένα γενικότερο σχόλιο τώρα. Η σημαντική ηγετική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προάθεση των στόχων για το κλίμα. Είναι σημαντική και Χαίρομαι για το γεγονό ότι η πολιτική αυτή μας ανοίγει τη δυνατότητα να προωθήσουμε και την βιώσιμη ανάπτυξη. Παλαιότερα στη κοινωνία των πολιτών είχε την τάση να κατακρίνει τον ΠΟΕ επειδή υποτίθεται ότι εκείνος ο ΠΟΕ δεν επέτρεπε την εφαρμογή ορισμένων ε, εθνικών ε, ή τοπικών πολιτικών. Πολιτικών οι οποίες, ε, στις οποίες είχαν καταλήξει τα κράτη μετά από πολύχρονες διαπραγματεύσεις, συζητήσεις που αντικοτόπτριζαν το πώς είχε εξελιχθεί η συζήτηση στις χώρες αυτές. Νομίζω σήμερα τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα γιατί έχουμε νομολογία από το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ που διευκρινίζει ότι τα κράτη-μέλη του ΠΟΕ έχουν δικαίωμα να υιοθετούν εθνικές πολιτικές για ζητήματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία δημοσίων αγαθών, η προστασία του καταναλωτή ή οποιοδήποτε άλλον εύλογο στόχο. Στο προήμιο της Συμφωνίας του Μαρακές υπάρχει αναφορά στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, στην προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος. Με βάση αυτό το προήμιο ερμηνεύουμε το άρθρο 20 του ΓΚΑΤ που περιγράφει τις ε, εξαιρέσεις που μπορεί να... που είναι η ρήτρα εξαίρεσης. Τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τέτοιες... να πολιτικές αποφάσεις, ακόμα και αν αυτές οδηγούν σε περιορισμούς. Βέβαια, οι περιορισμοί αυτοί θα πρέπει να είναι αναλογικοί, να μην είναι πιο περιοριστικοί από όσο χρειάζεται, να μην δημιουργούν διακρίσεις υπέρ ε, ε, εθνικών προϊόντων ή εναντίον προϊόντων άλλων χωρών και θα πρέπει να μην είναι ουσιαστικά ένα καμουφλαρισμένο προστατευτικό μέτρο σε αυτό το πλαίσιο, από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να ακολουθεί όποια πολιτική επιθυμεί. Η προστασία του περιβάλλοντος αντιμετωπίζεται επίσης και στην δομή του ΠΟΕ. Οι ιδρυτές του ΠΟΕ θεώρησαν ότι ήταν σημαντικό να δημιουργηθεί και μια επιτροπή για το ε, εμπόριο και το περιβάλλον. Εδώ είναι που συζητούνται ε, τέτοια θέματα όπως η κυκλική οικονομία, ή επίσης τα προβλήματα που δημιουργεί η αλόγιστη χρήση πλαστικού. Υπό την αιγίδα, την ηγεσία μάλλον της Γαλλικής Προεδρίας, τα μέλη υπο την ηγιδα την ηγεσια μαλλον της Επιτροπής έχουν συζητήσει τέτοια θέματα στην Υπουργική Διάσκεψη του Σοζούτα. Με ένα θέμα για το οποίο συχνά μας υποβάλλονται ερωτήματα είναι η τα τέλη για την, τον τρόπο μάλλον προσαρμογής στη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό δεν είναι ε, ένα πρόβλημα που αφορά μόνο την Ευρώπη. Είναι ένα πρόβλημα που έχει σχέση με το πώς συλλέγονται τα στοιχεία, για το πώς γίνονται οι υπολογισμοί. Το γεγονός ότι ε, η χώρα η οποία ε, δημιουργεί την μόλυνση θα μπορούσε να ε, ε, υποβάλει στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι έχει εθνικά προγράμματα αντισταθμιστικά. Έχει συμβεί κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Όμως δεν μπορείτε να περιμένετε από τον ΠΟΕ εκ των προτέρων να γνωμοδοτήσει για την νομιμότητα ή όχι οποιοδήποτε συστήματος υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε. Θέτετε πολλά ενδιαφερόντα ζητήματα, λέει η πρόεδρος, στον Ιστρία μάλλον. Τελευταίος μας, ε, ο ο κύριος Μάρκ Μάι. Τι πιστεύει λοιπόν η κοινωνία των πολιτών. Yeah, thank you, um, for inviting me here. Ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ. Στο προηγούμενο πάνελ καθόμουν στην αίθουσα και σκεφτόμουν εμείς ε, προερχόμαστε από ένα συνασπισμό ΜΚΟ για την ανάπτυξη. Όλα αυτά τα λειτουργικά προβλήματα που συζητάμε εδώ, αυτά με απασχολήσαν. Καλώς επιστρέψαμε τώρα στον τρίτο κόσμο. Οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη είναι πολύ βασικά πράγματα. Ε, φτώχεια, πείνα, ε, πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, στην υγεία και ούτω καθεξής. Και βασικά πράγματα. Και τι κάνει το εμπόριο για αυτά τα πολύ βασικά ουσιαστικά πράγματα. Αυτό είναι το ερώτημα. Και αυτό που ακούμε συχνά. Και αν δείτε ποια είναι η σχέση, όπως περιγράφεται μεταξύ εμπορίου και στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, βλέπουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι το εμπόριο συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και συνεπώς εισοδήματα, χρηματοδοτεί λοιπόν τα πάντα. χρηματοδοτεί όλου του στόχου βέσιμη ανάπτυξη και οτιδήποτε συμβόλαιο διότι το εμπόριο κινεί τον κόσμο. Έτσι λέμε. Το οποίο κατά συνέπεια σημαίνει ότι το εμπόριο είναι μια χαρά. Τα πάμε μια χαρά αφού δημιουργούμε αγορέ, πλούτο, υποστηρίζουμε του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη κατά συνέπεια και δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ωστόσο, αυτό που συχνά ξεχνάμε είναι ότι αυτή η σχέση μεταξύ του ανοίγματο αγορά και της ανάπτυξης και των εισοδημάτων δεν είναι και τόσο καθαρή. Έχουμε και ανεπτυγμένες αγορές χωρίς ανάπτυξη της οικονομίας και αυτοί που αποφελούνται είναι αυτοί που ήδη είναι πολύ εύποροι. Οπότε αυτή η μετακύληση στα εκατότερα στρώματα είναι μεγάλο θέμα συζήτησης. Αλλά αυτή είναι η λογική με στις άκρες. Και αυτό που βλέπετε τώρα, ε, βλέπετε αυτόν τον άνθρωπο στο Λευκό Οίκο, τους εμπορικούς πολέμους, ε, κάτι που επηρεάζει άμεσα την οικονομική ανάπτυξη παντού. Να δούμε τι σημερινέ συμφωνίε ελευθερών συναλλαγών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και συζητήσαμε πρόσφατα για τη ΣΕΙΤΑ πολύ. Η αξιολόγηση τη ΣΕΤΑ αναφέρεται σε ανάπτυξη 0,05 έως 0,06% ελάχιστη δηλαδή σε σχέση με το μέγεθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που βλέπουμε αντιθέτως είναι μεγάλη αύξηση του εμπόριου αλλά ελάχιστη οικονομική ανάπτυξη τι κάνει δηλαδή αυτή η ανάπτυξη του εμπορίου τελικά. Στέλνουμε γάλα στους Καναδούς, ε, αντικαθιστώντας το δικό τους γάλα, αυτοί στέλνουν κρέα σε εμά και εμείς έχουμε ένα σωρό κρέατα, αντικαθιστούν τα δικά μας. Πολύ εμπόριο δηλαδή που τρέχει, αλλά η ανάπτυξη. Πώς ε, συμβάλλει το εμπόριο στην ανάπτυξη. Και αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Πρέπει να δούμε δηλαδή αυτές τις διαδικασίες. Αυτός είναι ένας τρόπος ε, να δούμε τη σχέση μεταξύ εμπορίου και των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη. Το δεύτερο ερώτημα είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι εμπορικοί στόχοι μεταξύ των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε από του 69 στοχου 7 7-9 που σχετίζονται με το εμπόριο. Το, το 8 είναι το εμπόριο, η προώθηση, η προσέλκυση επενδύσεων επίση περιλαμβάνεται σε αυτούς. είναι συζητήσιμο πώς πραγματικά είναι αλλά αν τους δείτε πιο συγκεκριμένα αυτούς τους συγκεκριμένους στόχους δεν δείχνουν και πολύ καλά αποτελέσματα. Ένα από τους σημαντικούς στόχους, ο 17-10, ανοιχτό και ισότιμο παγκόσμιο σύστημα και επιτυχής ολοκλήρωση του γύρου της Ντουάλα. Το Σεπτεμβρίο του 2015 ε, υιοθετήθηκε το θεματολόγιο 2030 και το Σεπτέμβριο του 2015 στο Ναϊρόμπι. Οι πλούσιες χώρες προσπάθησαν να κάνουν εξοκύλιο γύρω στις Δόχα αφού δεσμεύτηκαν να επιτύχει ο γύρος της Δόχα. Μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση ο γύρος της Δόχα τελικά δεν επιβεβαιώθηκε, ακόμα ε, είναι σε κόμμα μάλλον. Uh, αυτό ήταν ένα από τους συγκεκριμένους στόχους ε, μεταξύ των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη. Υπάρχει και ένα άλλο για το διπλασιασμό των εξαγών των LDC μέχρι το 2020 των λιγότερων αναπτυγμένων χωρών. Δηλαδή αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Είμαστε στο 2020. Δεν ξέρω ποιο ήταν υπεύθυνο για κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό είναι ένα από του στόχου που δεν θα γίνει πραγματικότητα. Η αναφορά στην πρόσβαση σε φάρμακα και η απόφαση TRIPS ε, που ελήφθη στην Τόχα πριν πολύ καιρό. Ακόμα γίνεται αναφορά σε αυτό. Δεν χρησιμοποιείται ιδιαίτερα, αλλά στο διάμεσο, Ενώ αυτή η απόφαση εξακολουθεί να υπάρχει, οι φαρμακοβιομηχανίες ε, επινόησαν την προστασία των δεδομένων και την αποκλειστικότητα των δεδομένων που επεκτείνονται σε πολλά χρόνια με μείωση την πρόσβαση στα φάρμακα. Ω αποτέλεσμα και δεν ξέρω στο πλαίσιο τώρα των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη, αν γίνονται επιπλέον προσπάθειε για να φελτιωθεί αυτή. Υπάρχει το αδασμολόγητο ε, η αδασμολόγητη πτυχή στην εμπορική πολιτική χωρίς ποσοστώσεις που μετά από την διάσκεψη για τις LTC, για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, ελήφθη αυτή η απόφαση, αλλά πολλές χώρες δεν έχουν ακόμα φτάσει σε αυτό και δεν έχουν συμφωνήσει ούτε οι Αμερικανοί πολύ πριν έρθει ο Τραμπ στα πράγματα στη Βόσιγκτον, Η ειδική διαφοροποιημένη ε, μεταχείριση είναι από του συγκεκριμένους στόχους βιώσιμη ανάπτυξη. Ακόμα συζητείται σήμερα και μετά έχουμε το θέμα της αλίας. Πολύ δύσκολη συζήτηση, όπως θα ακούσατε και δεν είναι βέβαιο κατά πόσο θα επιτύχει, θα φέρει αποτελέσματα. Αυτό δείχνει ότι είναι δύσκολο να εντάξουμε συγκεκριμένους στόχους βιώσιμης ε, ανάπτυξη στην εμπορική πολιτική. Πώ συμβάλλει λοιπόν η εμπορική πολιτική σε αυτού, δεν είναι αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα είναι πώ μπορούμε να κάνουμε πιο βιώσιμη την εμπορική πολιτική, ούτω ώστε να ενταχθούν όλο και περισσότερο από αυτού του στόχου ε, στη χάραξη αποφάσεων εμπορική πολιτική. Και εκεί ακριβώ αυτό είναι που θα έπρεπε να γίνει. Διότι η Ατζέντα 2030 το λέει καθαρά. Οι 17 στόχοι και οι 169 επιμέρους στόχοι είναι μαζί και όλα αυτά θα πρέπει να συμβάλλουν σε όλους αυτούς τους στόχους από κοινού, στο βορρά, στο νότο και σε όλες τις διαφορετικές πολιτικές. Και η εμπορική πολιτική λοιπόν θα πρέπει να κάνει προσπάθειες να συμβάλλει σε όλα αυτά, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι ορατές. Και αυτό που λέμε εμείς είναι ότι εντάξει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πρέπει να γίνουν αξιολογήσεις ε, ε, βιωσιμότητας ε, για να δούμε κατά πόσο δημιουργείται βλάβη και το πώς γίνονται όλα αυτά είναι συζητήσιμο αλλά επίσης θα πρέπει να διαβεβαιώνουμε όχι μόνο ότι δεν είναι επιβλαβής αλλά ότι δεν αφήνουν κανέναν πίσω. Θα θέλαμε δηλαδή η ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική στο επίπεδο τη διαπραγμάτευση με αναπτυσσόμενε χώρες θα λαμβάνει υπόψη του 169 στόχου. και θα προβληματίζεται για το τι μπορεί να σημαίνει η εμπορική πολιτική για, όσον αφορά τους τάδε στόχους. Για πολλούς στόχους η εμπορική πολιτική δεν μπορεί να κάνει πολλά, αλλά για άλλους, πολλοί αριθμούς, στόχους ε, μπορεί κανείς να αναρωτηθεί. Η φτώχεια, η ανισότητα, η πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες, τι μπορεί να κάνει η εμπορική πολιτική για να βοηθήσει εκεί ή τι δεν πρέπει να κάνει. Γιατί δεν πρέπει να υπονομεύει φυσικά τις ε, κρατικές υπηρεσίες ε, που έχουν συσταθεί για αυτό το σκοπό. Για να σα δώσω ένα παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται με την Ινδονησία. Τι μπορεί να σημαίνουν αυτέ ε, οι διαπραγματεύσει για του ψαράδε. Ενδιαφέρον ερώτημα. Τι μπορεί να κάνει μια τέτοια συμφωνία. Ξέρουμε ότι οι ψαράδε ε, υποφέρουν λόγω των εχθεοκαλλιεργιών ε, για την καλλιέργεια γαρίδων. για την ε, που ρηπαίνει τα ύδατα, υποφέρουν αυτοί γιατί δεν πουλάνε αρκετά, τεράστια ξενοδοχειακές μονάδες χτίζονται και διώχνουν τους ψαράδες, ε, τεράστια αλλιευτικά σκάφη τους ανταγωνίζονται. Τι μπορεί λοιπόν να προσφέρει η εμπορική συμφωνία στους απλούς ψαράδες και να μην μιλάμε απλά για συνοδευτικά μέτρα. Να τους μάθουμε να, χτίζουν, να κατασκευάζουν πράγματα που θα μπορούν να πουλούν ας πούμε στις παραλίες σε τουρίστες όπου χτίστηκαν αυτά τα ξενοδοχεία. Να βρούμε τρόπους να επιβιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Επίσης, στην εμπορική πολιτική θα πρέπει να δούμε και πιο πέρα από αυτά. Η κλιματική αλλαγή δεν ήταν τόσο ορατή πριν πέντε χρόνια όπως είναι σήμερα σήμερα αποτελεί το βασικότερο πρόβλημα, η κλιματική αλλαγή αλλά και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος που συνεχίζονται το τεράστιο αποτύπωμα που έχουμε εμείς ε, στην Ευρώπη 1,7% 1,7 ε, φορές συγγνώμη πάντα κάνω λάθος με αυτό καταναλώνουμε 1,7 ε, φορές περισσότερα από ό,τι παράγουμε εμείς ήδη βασιζόμαστε δηλαδή σε μεγάλο βαθμό στον υπόλοιπο κόσμο και αν όλοι κάνουν το ίδιο έτσι όπως εμείς θα χρειαστούμε και άλλους πλανήτες εκτός από το δικό μας. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πιο πέρα από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να οργανώσουμε τη μετάβαση σε λιγότερες εκπομπές, σε μια κυκλική οικονομία. Για να το επιτύχουμε αυτό, Πρέπει να αναθεωρήσουμε τις 40 ε, συμφωνίες που έχει με αυτές τις 70 χώρες Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, στην κυκλική οικονομία υπάρχουν εταιρείε που εμπλέκονται στην ανακύκλωση. Λένε δηλαδή πάμε και παίρνουμε ό,τι περισσεύει από μια παραγωγή και μετά ε, εξάγουμε τα απο, απορρίμματα αυτών των ε, παραγωγών, αλλά εμεί θέλουμε τα κρατάμε εδώ να τα κυκλώνουμε. Αλλά αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε απαγορεύσει εξαγωγών. Πρέπει να ξαναπάμε πίσω δηλαδή και να ξαναδούμε τι συμφωνίε ε, που υπάρχουν για τι εξαγωγέ, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι τα απόβλητα θα παραμένουν στην Ευρώπη. Αν πάμε δηλαδή να δούμε πιο ανοιχτό αλλά πιο πέρα από αυτά που έχουμε σήμερα και από τι σημερινέ μα ανάγκε, τότε μπορεί να επινοήσουμε νέου ε, τρόπου εμπορική πολιτική. Είναι τεράστια η θεματολογία. Λέει η συντονίστρια, θα πρέπει να επιταχύνουμε. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στους βουλευτές που το επιθυμούν. Έχω πρώτα τον Κρίστοφ Χάνσεν πρώτο. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τους τρεις ομιλητές έχω κάποια σχόλια και ερωτήσεις. Ε, ευχαριστώ κύριε Καρλ Μπράουνερ για την εισήγησή σας, αλλά και για τις ανησυχίες που αναφέρατε για την Αλία. Είχαμε την ευκαιρία να ε, συναντηθούμε στις αρχές του Δεκεμβρίου στη Γενέβη. Εγώ είμαι από το Λεξεμβούργο που δεν είναι χώρα της Αλίας, γιατί δεν έχουμε πρόσβαση στη θάλασσα ως χώρα. Ωστόσο ανησυχώ για το ποια είναι η θέση στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο σε σχέση με το EMFF και Μιλάμε για 6 δις, οπότε πολλοί κόσμος λέει δεν είναι πολλά τα χρήματα, αλλά η ζημιά που μπορεί να κάνουν αυτά τα χρήματα μπορεί να είναι μεγάλη. Και είναι πολύ ε, τρομακτικό αυτό. Έχω μελετήσει αυτή την υπόθεση και έχω την αίσθηση ότι εμείς παραβαίνουμε ο στόχος του 40,6 όσον αφορά για τις περιβαλλοντικά βλαβερές επιδοτήσεις και πρέπει να προσέξουμε να έρθουμε σε επαφή με άλλες αντιπροσωπείες στη Γενέβη όπως ο πρέσβης την που έθιξε αυτό το θέμα. Δηλαδή αν θέλουμε να δούμε μελλοντικέ διαμάχες ή διαπραγματεύσεις θα πρέπει εδώ να προσέξουμε πάρα πολύ τι κάνουμε. Αλλά δεν μιλάμε μόνο για την αλληλεία και έναν στόχο Έχουμε και τον στόχο 13 για την κλιματική δράση. Εκεί είχα την ευκαιρία να συμμετέχω στη Μαδρίτη στη διάσκεψη για το κλίμα με την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου. Είχαμε και πολλές αντιπροσωπείες τρίτων χωρών εκεί. Ας πούμε ρώτησα την Ιαπωνέζικη αντιπροσωπεία γιατί ήμουν σκιώδη στη ΣΥΝΤΑ για την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιαπωνίας για την ελεύθερη, ελεύθερη ε, και τους ρώτησαν αν έχουν ε, τις ίδιες δεσμεύσεις ε, όπως για τους στόχους του Παρισιού όταν διαπραγματευτήκατε την Διατλαντική Συμφωνία είδα τους δύο συνομιλητές να μιλάνε να κοιτούνται παραξενεμένοι γιατί δεν περίμεναν ότι θα προκύψει αυτό. Καλό θα ήταν να υπάρχει λοιπόν ισότιμο πεδίο ανάμεσα σε τρίτες χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά έχω την εντύπωση πως υπάρχει κάτι που δεν αναφέρεται συχνά. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ασχολούνται με το εμπόριο και τι εμπορικέ διαπραγματεύσει δεν επικοινωνούν με του συναδέλφου του που ασχολούνται με το κλίμα και το περιβάλλον. Σήμερα το πρωί πήραμε πράσινο φως, ε, μάλλον δώσαμε το πράσινο φως για την εταιρική σχέση με το Βιετνάμ. Και εκεί έχουμε ένα κεφάλαιο για το εμπόριο και ζητάμε να συσταθεί μια κοινή επιτροπή για να επιβλέπει την εφαρμογή της ε, συμφωνίας αυτή ε, με το Βιετνάμ. Ε, θεωρείτε ότι μπορεί αυτό να αποτελέσει παράδειγμα για άλλες εμπορικές συμφωνίες με άλλους εταίρους. Σας ευχαριστώ πολύ. Κατλίν Φαν Μπρέμπτ. Όχι, ναι, καλά το είπατε το όνομά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, υπάρχουν τόσο πολλά για συζήτηση και με εμπνεύσατε πάρα πολύ, αλλά έχω την εντύπωση πως η συντονίστριά μας είναι ε, πολύ σκληρή, όπως και ο πρόεδρος της Επιτροπής μας, που είναι ο συνήθες ε, συντονιστής μας. Θα κάνω μια γενική παρατήρηση. Εγώ είμαι νέα σε αυτή την Επιτροπή και νομίζω πως ε, μία από τις πρώτες συνεδριάσεις το ακούσαμε από την πρώην ε, Επίτροπο για το εμπόριο Μόλμστρομ που είπε το περίφημο ε, το εμπόριο δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα του κόσμου. Και πολλοί έκτοτε έχουν επαναλάβει αυτή τη φράση. Αν και δεν είναι ότι διαφωνώ απόλυτα, έχει γίνει ένα ε, τροπάριο που όμως δυστυχώς δεν είναι αυτός ο τρόπος για να προχωρήσουμε όταν αναφέρθηκε στην κλιματική πολιτική, είπε και σωστά ότι δεν είναι το πώς θα βάλουμε την κλιματική πολιτική στο, εμπόριο, αλλά το εμπόριο θα αλλάξει πολύ λόγω των κλιματικών αλλαγών και αυτό θα πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Χρειαζόμαστε ένα συγκεκριμένο καθεστώς για τους κλιματικούς πρόσφυγες, ας πούμε, ενώ ξέρουμε ότι υπάρχει διασύνδεση με το κλίμα και το τι συμβαίνει στο κλίμα το εμπόριο, την οικονομία και ούτω καθεξής. Και αυτή είναι δική μας ευθύνη, σε αυτήν εδώ την Επιτροπή, να δούμε αυτή την σύνδεση εντάξει, αυτών των τομέων. Είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε και να συνεργαστούμε και με άλλες επιτροπές. Γιατί εργαζόμαστε λίγο απομονωμένα. Πρέπει να ανοίξουμε και να συνεργαστούμε. Θα μιλήσω για τη στρατηγική για την Αφρική, γιατί είναι ένα θέμα σημαντικό. Και το εμπόριο είναι μεγάλο κομμάτι. Η αναπτύξη είναι στο ε, προσκήνιο, αλλά και το εμπόριο είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ έχω μια ερώτηση προς τους πανελίστες. Πώς το βλέπουν να μας συμβουλέψουν, γιατί τώρα ξεκινάμε τις συζητήσεις. Να, τώρα εξετάζουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε μεγάλες επικρίσεις για τη ΣΕΠΑ και το πώς αντιμετωπίζουμε την Αφρική είναι πως δεν επιτρέπουμε στην Αφρική να αποκτήσει μια εσωτερική αγορά όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή να έχουν μια αξία, μια λυσίδα αξία. Ας πούμε η σοκολάτα είναι πολύ καλό παράδειγμα. Έχουν πολλές εξαγωγές από τη Δυτική Αφρική προς ε, τον υπόλοιπο κόσμο και στην Ευρώπη. Και ενώ ταυτόχρονα η παραγωγή σοκολάτα στην Αίγυπτο, ας πούμε, η, η, η Αίγυπτος, ας πούμε, δεν παίρνει σοκολάτα από την Αφρική. Είναι ένα απλό παράδειγμα και υπάρχουν πάρα πολλά άλλα τέτοια παραδείγματα. Όταν βλέπουμε την ανάπτυξη, την, την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης, τι πρέπει να αλλάξει στην εμπορική πολιτική της Ευρώπης με την Αφρική. Μπορείτε να μας δώσετε πέντε τρόπους να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Και κάτι ακόμα. Έχουμε το νέο πράσινο σύμφωνο. Εγώ πιστεύω πως είναι ο τρόπος για να προχωρήσει η Ευρώπη, αλλά δεν θα πετύχει ποτέ νομίζω εάν δεν ενταχθεί αυτό, να δεν συνοδοματωθεί στην εμπορική μας πολιτική, όχι μόνο για, την, για τον άνθρακα. Ναι, εντάξει, αυτό πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να γίνουν και περισσότερα. τα κεφάλαια TSD ας πούμε είναι πολύ σημαντικό που είναι εκεί ε, που υπάρχουν καν αλλά δεν περιλαμβάνουν κυρώσεις δεν... Ε, συγγνώμη που αυτά είχα να πω. Η Άννα Καβατσίνη είναι η επόμενη. Σας ευχαριστώ και από τη δική μου την πλευρά για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Χαίρομαι επίση που ξαναβλέπω παλιού συναδέλφους, σε σας αναφέρομαι Ιζαμπέλ. Θα συνεχίσω τη σκέψη της κυρίας Φαμπρέντ. Έχουμε το πράσινο σύμφωνο και επίσης ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμα για το πράσινο σύμφωνο έχουμε αποφασίσει ότι θα συνδέουμε τις εμπορικές μας συμφωνίες με περιβαλλοντικούς στόχους και πιο συγκεκριμένα με στόχους για την συμφωνία το, της, για την κλιματική αλλαγή των Παρισίων, το οποίο σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη αποφασίσει να αξιοποιήσει την εμπορική πολιτική για την προώθηση των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη. Όμω, συνεχίζουμε να έχουμε μια έλλειψη και χρειαζόμαστε συγκεκριμένε προτάσει για το πώ μπορεί αυτό να συμβαίνει γενικότερα. Δηλαδή, υπάρχουν άλλε μεταρρυθμίσει που πιθανώ θα μπορούσαμε να επιφέρουμε στους κανόνες του ΠΟΕ ή για παράδειγμα οι προτάσεις του Μακρόν για ε, ε, ε, άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη των ομιλητών μας για άλλους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί η εμπορική πολιτική για το περιβάλλον. Ο επόμενο ομιλητή ο κύριο Σόλτ. Ευχαριστώ, σα ευχαριστούμε για τι ενδιαφέρουσε παρουσιάσει. θα έλεγα ότι στις γενικές γραμμές υπάρχει συμφωνία. Και αναφερόμαστε στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης με πάνω κάτω τον κοινό τρόπο. Αναφέρθηκε για ένα συγκεκριμένο παράδειγμα η Αλία. Όμως, κατά το παρελθόν έχουμε πει ότι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να θεωρούνται ως μια ε, μέτρο ε, της επιτυχίας, ένα εγκάρσιο μέτρο της επιτυχίας όλων των πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο τη εμπορική πολιτική τη. Και υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της Γινέβης κάποιοι πράσινοι στόχοι, πέντε αρχές μάλλον, πέντε αρχές, ανάμεσα στις οποίες η προώθηση της πολυμέρειας. Και η τέταρτη ήταν ότι οι διεθνείς κανόνες θα πρέπει να δημιουργούνται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να προλαμβάνουν ε, καταστροφτικές μονομερείς ενέργειες οι οποίες να αποτρέπουν από άλλα κράτη, να, οι οποίες να μπορούν να οδηγήσουν σε άλλα κράτη να μην έχουν τη δυνατότητα να ε, πετύχουν τους στόχους τους. Το οποίο σημαίνει ότι αυτό και αυτές τις πέντε αρχές τις έχει ήδη αποδεχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στις διαπραγματεύσεις της με άλλες τρίτες χώρες. Και φυσικά αυτό μπορεί κάποιος να το επικαλεστεί. Δώστε μου λοιπόν ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε την οικονομική πολιτική και την εμπορική πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση. Και έρχεται το ερώτημά μου προς τον κύριο Μαές. Ε, γιατί εσείς μιλήσατε για τις εξαγωγές και είπατε ότι πρέπει να επανέλθουμε σε μια προτεραιά κατάσταση. Εσείς τι πιστεύετε λοιπόν, πώς μπορεί αυτό να γίνει συμβατό με τη σημερινή κατάσταση. Πιστεύετε ότι είναι σωστή η προσπάθεια που γίνεται να οργανώσουμε την διμερή ή πολυμερή ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών ή μήπως θα λέγατε ότι πρέπει να επανέλθουμε στις βασικές αρχές των υποχρεώσεων που θεσπίζουν το Ηνωμένα Έθνη, άρα να υπάρχουν όλο και περισσότερες συμφωνίες συνεργασίας. Και αυτή η συζήτηση μας ξαναγυρνά στην ουσία της ε, μιας εμπορικής πολιτικής. Κυρία Τσάνς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Δύο θέματα θα ήθελα να θίξω. Πρώτον προς την κυρία Τιουγό. Χαίρομαι που επενθυμίσατε ότι η οικονομία πρέπει να λειτουργεί προ όφελο των πολιτών, προ όφελο των ανθρώπων και όχι το αντίστροφο. Το είπατε ξεκάθαρο. Στον προηγούμενο γύρο ερωτήσεων υπήρξαν κάποιοι βουλευτές από άλλε πολιτικέ ομάδες που ε, με ε, εντυπωσίασαν αρνητικά επειδή είχαν μια απλοποιημένη ε, μανιχαϊστική προσέγγιση, δηλαδή ότι μπορεί κανείς να είναι υπέρ ή κατά του εμπορίου. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί κάποιο να είναι υπέρ, ε, μάλλον ότι είναι υπεραπλουστευτικό το να, το να είναι κανείς υπέρ του εμπορίου σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι το ερώτημα εάν περισσότερο ή λιγότερο εμπόριο θέλουμε. Το ερώτημα είναι ποιας ποιότητας είναι αυτό το διεθνές εμπόριο. Και ένα πρόβλημα είναι ότι μόνο ποσοτικούς δείκτες χρησιμοποιούμε για να αξιολογήσουμε το διεθνές εμπόριο και ίσως ένα πρόβλημα να είναι ακριβώς αυτό, ότι δεν χρειαζόμασταν και ποιοτικού δείκτες. Και αυτό είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα που θα ήθελα να θέσω σε ολόκληρο το πάνελ. Πώς μπορούμε να απομακρυνθούμε από αυτήν την υπεραπλουστευτική μεθοδολογία που βασίζεται μόνο σε ποσοτικούς δείκτες και να πάμε όλο και περισσότερο σε δείκτες οι οποίοι να αντικατοπτρίζουν την κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση του, των επιπτώσεων του διεθνούς εμπορίου. Να μην κοιτάμε δηλαδή μόνο την αύξηση του ρυθμού των εξαγωγών του ΑΕΠ. Το δεύτερο. Προ τον εκπρόσωπο του ΠΟΕ, βεβαίω συμμερίζομαι τι ανησυχίε σα για την αλληλεία αλλά με παραξένεψαν οι παρέμβασή σας, γιατί ουσιαστικά μας είπατε ότι εντάξει, βασικά δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα η λειτουργία του ΠΟΑ για, για τη βιώσιμη ανάπτυξη, γιατί υπάρχει ένα πεδίο ε, ελιγμών. Ε, η δικιά μου εμπειρία και οι δικές μου γνώσεις δείχνουν ότι θα μπορούσε κανείς να είναι πολύ πιο φιλόδοξος. Ότι στην πραγματικότητα χρειάζονται επιγόντως μεταρρυθμίσεις στον ΠΟΕ. Μια και λοιπόν τουλάχιστον αναγνωρίστηκε σε διεθνέ επίπεδο η ύπαρξη μια παγκόσμια κλιματική κρίση, κάτι που δεν συνέβαινε πριν από πέντε χρόνια. Μήπω μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό για να πάμε ένα βήμα περιπέρα. Όχι απλώ να λέμε ότι είναι επαρκέ να μην βλάπτει ο ΠΟΕ το περιβάλλον, αλλά πώς θα μπορέσουμε να τον μεταρρυθμίσουμε έτσι ώστε να συνεισφέρει στο περιβάλλον. Και, κάτι, και, αυτή η, οποιαδήποτε ιδέα μπορείτε να μας δώσετε προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν καλοδεχούμενη. αυτό συνδέεται και με την ερώτηση της συναδέλφου Άννα προηγουμένω. Η κυρία Πινιέρο, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους τους ε, συμμετέχοντες. Εγώ ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια σύντομη σκέψη. Συζητούμε πολύ για το εάν θέλουμε ή όχι εμπόριο. Κανένας δεν είναι ε, ε, διατεθειμένος να αποφασίσει να πάψει να χρησιμοποιεί τα κινητό του, την ε, ε, επικοινωνία, τα να μην έχει τρόφιμα. Επομένως, με αυτή την έννοια το εμπόριο το χρειαζόμαστε. Το ζήτημα όμως είναι άλλο. Υπό ποιε συνθήκες παράγονται αυτά τα αγαθά και αυτές οι υπηρεσίες που μετά εμπορευόμαστε. Αυτή είναι η ουσία της συζήτησης. Όχι να συζητάμε θέλουμε ή δεν θέλουμε εμπόριο. Και οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης βασίζονται στην φιλοσοφία ότι αν η ανάπτυξη δεν είναι βιώσιμη, δεν είναι ανάπτυξη. Και η κλιματική αλλαγή έχει έρθει πλήρως στο προσκήνιο των συζητήσεών μας. Όμως, δεν είναι ζήτημα ε, βιωσιμο... Η βιωσιμότητα μάλλον δεν είναι μόνο ζήτημα περιβάλλοντος, προστασίας του περιβάλλοντος. Υπάρχει και η κοινωνική βιωσιμότητα, η βιωσιμότητα ως προς τα... το σεβασμό των εργατικών δικαιωμάτων. Και εγώ θα πρόσθετα επίση και την ισότητα των δύο φύλων θα έπρεπε να το δούμε και αυτό το πρόβλημα ε, ως ζήτημα βιωσιμότητας, γιατί θα πρέπει όλος ο πληθυσμός να έχει τις ίδιες ευκαιρίες, είναι και αυτό θεμελιώδης σημασία. Και εξάλλου υπάρχουν πολλές μελέτες που αποδεικνύουν ότι ο ΠΟΕ θα μπορούσε και θα έπρεπε να κάνει πολλά περισσότερα για αυτούς τους στόχους είναι θέματα τα οποία τα συζητούμε ε, εδώ και πάρα πολύ καιρό και σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Και θα ήθελα να απευθύνω αυτό το ερώτημα στον κύριο Μπράουν, λοιπόν, για συγκεκριμένα για τα προβλήματα αυτά τι κάνει ο ΠΟΕ. Όσον αφορά τώρα τα ανθρώπινα δικαιώματα, λέμε ότι είναι απολύτω απαραίτητο να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά δικαιώματα, τα εργατικά δικαιώματα, να μην υπάρχει εκμετάλλευση στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Μια σημαντική πρωτοβουλία έχουν αναλάβει τα Ηνωμένα Έθνη για να εξασφαλιστεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις επιχειρήσεις. Και βεβαίως ξέρουμε ότι ακόμα δεν έχει υπάρξει συμφωνία για το θέμα αυτό στο, στο Συμβούλιο. Είναι γνωστό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει την υποστήριξή του σε αυτή την πρωτοβουλία. Όμως όλοι εμείς που θέλουμε να προωθήσουμε την βιώσιμη ανάπτυξη, πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη δημιουργία μιας διεθνούς συνθήκης νομικά δεσμευτικής, έτσι ώστε να απαιτείται από τις επιχειρήσεις να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δικαίωμα στη ζωή και άλλα εξαιρετικά σημαντικά δικαιώματα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πούν οι ομιλητέ μα τι πιστεύουν για αυτό, τι πιστεύουν για τη δημιουργία μια τέτοια νομικά δεσμευτική ε, συνθήκη. Και τέλο. Ε, εμείς, ε, εγώ θα ήθελα να ακούσω από εσάς τι περιμένετε από εμά, τι περιμένετε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει για να σα βοηθήσει στι διάφορε ιδέε που μα προτείνατε. Η κυρία Κάτσμπρο, είχα πει και νωρίτερα ότι είναι θετική μέρα για το εμπόριο. Είχαμε ένα θετικό αποτέλεσμα για τη συμφωνία με το Βιετνάμ σήμερα το πρωί και ένα εξαιρετικό πάνελ σήμερα το απόγευμα, ε, δεύτερο πάνελ. Έχω δύο ερωτήσεις. οι εποχές αλλάζουν. Και σήμερα συζητάμε το εμπόριο και τη βιωσιμότητα αντί εμπόριο ή βιωσιμότητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα, μεγάλη αλλαγή σε σχέση με πριν από 10 χρόνια πιστεύω. Ενίοτε εστιαζόμαστε φυσικά στην κλιματική αλλαγή, πράγμα που δεν είναι παράξενο δεδομένου του κατεπήγοντος της κατάστασης. Ωστόσο πιστεύω ότι είναι σημαντικό η προσέγγιση μας να είναι ολιστική προς την βιώσιμη ανάπτυξη και ειδικότερα όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Μερικές φορές πιστεύω ξεχνάμε τη βιοπικιλότητα, για παράδειγμα. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η δική σας σκέψη όσον αφορά μια πιο ολιστική προσέγγιση μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα μαζί παράλληλα. Γιατί αλλιώ εστιαζόμαστε σε ένα πράγμα τώρα και σε δέκα χρόνια θα πρέπει να ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Πώ θα μπορούσαμε να έχουμε μια τόσο ολιστική προσέγγιση. you, raised, uh, to the... Και θα κάνω και την ίδια ερώτηση και στο δικό σας πάνελ όπως έκανα και στο προηγούμενο πάνελ. Υπάρχει ένα θέμα που θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο και που με απασχολεί πολύ οι επιδοτήσεις στα ορεκτά καύσιμα που πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να ξεφορτωθούμε. Αλλά και πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο να βρω και άλλες ε, καθολικές ε, διαδικασίες ε, που έχουμε εντοπίσει και που έχουμε συμφωνήσει να βοηθήσουμε να εξαλείψουμε σιγά σιγά. Ποιες ιδέες έχετε εσείς. Επίσης συμφωνώ με τη συναδελφού. Καθόμαστε εδώ σε πάνελ. Μας παρουσιάζουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ιδέες αλλά ε, ας είμαστε ειλικρινείς, ε, ας μιλήσουμε ομά. Τι αναμένετε από τους πολιτικούς. Εμείς βρισκόμαστε εδώ για να βοηθήσουμε να επιτευχθούν αποτελέσματα και ίσως να μην εστιαζόμαστε στα σωστά πράγματα, διότι πέντε χρόνια είναι μικρό χρονικό διάστημα. Και το θέμα που συζητάμε αυτή τη στιγμή θα είναι πολύ πιο μακροχρόνιο. Οπότε σας παρακαλώ να κλείσουμε έτσι με απόλυτη ειλικρίνεια το σεμινάριο αυτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είμαι βέβαιο ότι θα γίνει έτσι. Να προτείνω, Καλ Μπράουνερ, ε, σας απίφθηναν συγκεκριμένες ερωτήσεις για τον ΜΠΟΕ. Αν θέλετε, αναφέρθηκαν στο διάστημα, στο φύλλο, στις επιδοτήσεις για την αλληλεία. Μπορείτε να απαντήσετε για αυτά και μετά Ιζαμπέλ να απαντήσετε ο... Ε, σε οποιαδήποτε ερώτηση φυσικά θέλετε. Ιζαμπέλ Τυρό, μετά υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις πολύ ενδιαφέρουσες θεωρώ για την ολιστική προσέγγιση, την προσέγγιση κατά τμήματα, διαφορετικές προτεραιότητες ε, και το πόσο ε, τα κεφάλαια των στόχων βιώσιμης ανάπτυξη είναι εφαρμόσιμα. Και οποιοδήποτε άλλο θέλει να σχολιάσει μπορεί ελεύθερα. Κύριε Μπράουνερ, να ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις ερωτήσεις. Κοιτάξτε, εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είστε αυτοί που εγγυάστε ότι η πολιτική αυτού του θεσμικού οργάνου θα βασίζεται σε αξίες. Εσείς είστε η τρανταχτή απόδειξη στις συμφωνίες που συνάπτετε εμπορικά ότι σας ενδιαφέρουν οι αξίες και έχετε και μηχανισμούς υλοποίησης. Δεν βλέπω λοιπόν να γίνεται κάτι λάθος. Εδώ στο Κοινοβούλιο ο κ. ρώτησε ε, ζήτησε να, να λαμβάνονται υπόψη στο βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις πολιτικές. Δεν μπορώ παρά να επικροτήσω τα όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό τον κλάδο, σε αυτό τον τομέα και πάντα υπάρχει φιλοδοξία να υπάρχει συμμόρφωση με τον ΠΟΕ. Για μένα λοιπόν, εμείς είμαστε οι καλοί μαθητές. Συνεχίστε έτσι. Άκουσα αυτά που είπε ο διπλανό μου και έχει δίκιο. Δεν ζούμε σε έναν ιδανικό τέλειο κόσμο. Πάντα μπορούν να γίνουν περισσότερα. Και συμφωνώ μαζί σα ότι η εμπορική πολιτική δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Έτσι έχουν τα πράγματα και θα πρέπει να ενθαρρυνθούμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι και άλλε πολιτικέ για να επιτύχουμε και άλλου στόχου. Τέθηκε το ζήτημα για το φύλλο. Ε, ουσιαστικά μετά από την Υπουργική Διάσκεψη των Buenos Aires, ε, ε, έχουμε μια κοινή ε, πρωτοβουλία για τις γυναίκες και το εμπόριο. Κάτι που εξελίχθηκε σε ένα θέμα το οποίο επίσης σχετίζεται με πολλά ζητήματα που συζητάμε σε πολλές διαφορετικές περιστάσεις γιατί αναγνωρίζεται φυσικά ότι οι γυναίκες παίζουν τεράστιο ρόλο για την ανάπτυξη. Έχω και εγώ τη δική μου προσωπική άποψη διέστηση ότι όλα τα προβλήματα του κόσμου θα, λυθούν, λύνονταν αν είχαμε περισσότερες γυναίκες ε, να απασχολούνται με αμοιβή. Η αμοιβόμενη εργασία των γυναικών είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Ευχαριστώ τον κύριο Χάνζεν που με υποστηρίζει για την εκκλησία μου όσον αφορά την Αλία. Και ναι, ε, δεν θέλω να ε, σας πάρω μονότερμα δώσουμε το λόγο και στους συναδέλφους. Απλά ήθελα να πω ότι προσπαθώ να σας εξηγήσω ότι ο ΠΟΕ δεν σας εμποδίζει να ακολουθείτε και να υλοποιείτε πολιτικές που εσείς θεωρείτε ότι αξίζουν. Τώρα τίθεται το ερώτημα του θα μπορούσε ο ΠΟΕ να υποστηρίζει πιο ενεργά ορισμένες πολιτικές. Το επίπεδο φιλοδοξίας ε, ορίζεται από την εθνική πολιτική, από τα κράτη-μέλη, στις εθνικές τους πολιτικές. Και μετά έτσι πρέπει να βρει κανεί τα σωστά εργαλεία για να μεταφέρει στο πολυμερέ σύστημα όλες αυτές τις φιλοδοξίες και σε συμφωνία φυσικά με τους επιμέρους εταίρους. Θα σταματήσω εδώ για να δώσω με το λόγο και στους συναδέλφους. Ευχαριστώ κύριε Ντουρό. Ευχαριστώ. Κάποια στοιχεία πρώτα για να απαντήσω και να δώσω στοιχεία στον κύριο Άνσεν. Ναι, εμπόριο και κλίμα δεν μιλούν μεταξύ του. Είναι δύο κόσμοι όπου οι διαπραγματευτέ δεν γνωρίζονται καν μεταξύ τους. Ε, διοργανώσαμε ένα ατελείο ε, για πρώτη φορά στη Γενέβη. Καλέσαμε 21 διαπραγματευτές σε κλίμα, εμπόριο, ε, ψηφιακός κόσμος. Τους φέραμε όλους μαζί κοντά και κάναμε μια συζήτηση για το κλίμα, εμπόριο και τα λοιπά Και ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί όντω αυτοί οι άνθρωποι δεν γνωρίζονται μεταξύ του και η κυρία τα έλεγε πως ε, κάποιες φορές και εδώ ε, δεν υπάρχει συνεργασία. Πρέπει να βελτιωθεί δηλαδή η, η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τμήματων. Και στον ΟΗΕ συμβαίνει το ίδιο. Για να συνδυαστεί το εμπόριο με το ε, κλίμα. Γιατί το έχουμε δει είναι αμφίδρομη η επιρροή. Το κλίμα επηρεάζει με θεαματικό τρόπο το εμπόριο, με καλό ή με κακό τρόπο ανάλογα πώς το βλέπει κανείς και τούμπαλιν. Να δούμε για την Αφρική. Ποιε είναι οι προτεραιότητες. Είναι αλήθεια ε, ότι η Αφρικανική Ένωση έκανε την επιλογή και αυτό κυρώθηκε από αρκετέ ε, αφρικανικέ χώρε να ξεκινήσουν μια ζώνη ελευθέρων συναλλαγών σε αφρικανική κλίμακα μπορεί να είναι πολύ καλή, εξαρτάται τι θα μπει εκεί και πώς μπορεί η Ένωση μαζί με άλλους, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορέσει να ε, ε, βοηθήσει ώστε να ε, λειτουργήσει μια τέτοια χώρα. Ας πούμε, αν μειωθούν οι δασμοί ανάμεσα στις περιφέρειες αφρικανικές, είναι πολύ περίπλοκο ακόμα και όταν κανείς θέλει να, να, να ε, ταξιδέψει στην Αφρική δεν, δεν υπάρχουν οριζόντιες συνδέσεις, όλα περνάνε από περιφερειακούς κόμβους. Α, περιφερειακή κλίμακα είναι πιο απλή, πιο εύκολη για τους πιο μικρούς παίκτες, ώστε να μπουν σε μια αλυσίδα αξία σε πιο ε, δίκαιη ε, για σε τεράστιες αλυσίδες ε, οι μικρότεροι είναι αυτοί που χάνουν συνήθως. Έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να δουλέψουμε πάνω σε αξίες που ε, προωθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο εμπορικού τύπου για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δηλαδή, αλλά για να υπάρξει μια λογική της αγοράς που να είναι ενδιαφέρουσα και να βοηθήσει στην, Αφρική, στην ανάπτυξη των χωρών της Αφρικής, ας πούμε, γεωγραφικές ενδείξεις. Θα μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε λοιπόν αναπτυξιακέ πολιτικέ τι αφρικανικέ που θα λαμβάνουν υπόψη τη γεωγραφική προέλευση. Πρόσφατα πήγα στο Περού, που δεν είναι βέβαια Αφρική, αλλά δουλεύουν πολύ για τη βιοπικιλότητα και πώ θα προστατεύσουν ταυτόχρονα τη βιοπικιλότητα, αλλά να έχουν ταυτόχρονα πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά για αυτό που ονομάζεται novel foods, ε, νέα τρόφιμα είναι πολύ δύσκολο, ε, δυσκολεύονται πολύ να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί οι κανόνες είναι εξαιρετικά αυστηροί. Δεν λέω να τους αλλάξουμε, αλλά πώς θα μπορούσαμε να δώσουμε κίνητρα και οικονομική δραστηριότητα που θα παρέχει κίνητρα στις χώρες που το χρειάζονται. Όσον αφορά τις περιφερειακές συναλλαγές, το τουρισμός επίσης είναι ένα στοιχείο ε, για βιώσιμη ανάπτυξη και οικονομική ανάπτυξη εάν τον σκεφτούμε με διαφορετικό τρόπο από ό,τι σήμερα. Μίλησα για την Καραϊβική πριν από λίγο γιατί δεν μπορούμε πάντοτε να λέμε πως ο τουρισμός λειτουργεί με βιώσιμο τρόπο. Κάθε άλλο μάλιστα. Και μετά για τη μετανάστευση όχι μόνο προς εμάς, αλλά και την ενδοαφρικανική μετανάστευση που είναι πολύ μεγάλη και που θα μπορούσε να δημιουργήσει πλούτο και ε, ανταλλαγές. Διαφοροποίηση της οικονομίας, ώστε να μπορέσουν οι αφρικανικές χώρες να διαφοροποιηθούν στις οικονομίες τους και να τους ενθαρρύνουμε για να μην εξαρτώνται από τα βασικά προϊόντα, για πράγμα που είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί όταν αλλάξουν τα προϊόντα, καταραίουν οι αγορές και οι συνέπειες είναι άμεσες. Τρίτο, τι μπορεί να κάνει η Κνουσέντη Ανκτάντ. Εμείς είμαστε μια διάσκεψη, δεν είμαστε πολιτικός φορέας, δεν είμαστε παίχτης. Έχουμε εντολή που μας ε, έρχεται από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο από τα κράτη ε, τα αναπτυσσόμενα, που είναι ας πούμε η ιστορία της ε, Ανκτάντη είναι ότι γεννήθηκε από τις αναπτυσσόμενες χώρες που ζήτησαν να τις βοηθήσουμε για να κάνουν εμπόριο με τρόπο που να βοηθά την ανάπτυξή τους. Δουλεύουμε μαζί τους αλλά με όλους. Βέβαια, με στη διάσκεψη υπάρχουν πολλώσεις, όπως και εδώ, ανάμεσα στους ε, G77, το οποίο και ο κύριος Μας, όπου η ατζέντα της ΔΟΧΑ ποτέ δεν ολοκληρώθηκε και δεν εφαρμόστηκε. Μεγάλη λοιπόν απόγνωση των χωρών που ξεχάστηκαν. Αυτή η ατζέντα δεν έχει εφαρμοστεί και άρα υπάρχει πόλωση ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες χώρες και τις άλλες. Δεν είναι εύκολο να αναζητηθούν νέες συμμαχίες για ορισμένα θέματα που θα επέτρεψαν να φύγουμε από την παραδοσιακή πόλαση, η οποία είναι κατανοητή μεν, αλλά οι νέες προκλήσεις ε, δεν σημαίνουν ότι οι παλιέ έχουν εξαλειφθεί. Τέλος. Business and Human Rights. Εδώ δεν ασχολείται ούτε η ΟΠΟΕ, ούτε η ε, Κνοσέντε είναι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έχει φτιάξει μια ομάδα εργασίας για να υποχρεώσει τις διεθνείς εταιρείες, τους διεθνείς όμιλους, τους ε, τις πολυεθνικές να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί όπου λειτουργούν. Δεν ξέρω τι θα βγει από αυτό. Ελπίζω πραγματικά πως κάτι θα βγει γιατί πιστεύω πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε νομικά επιχειρήματα αλλά πώς να εξηγήσουμε ότι οι πολυεθνικές ας πούμε εξαιρούνται από την εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ε, δεν υπάρχει λόγο να ισχύει κάτι τέτοιο. Όλοι θέλουμε να βοηθήσουμε. Εύκολο να το λέμε, αλλά λιγότερο εύκολο να γίνεται στην πράξη και οι διαπραγματεύσει δεν είναι ευπλέ, γιατί υπάρχει μεγάλη πόλωση. Ελπίζω πω οι διαπραγματευτέ θα βρουν τον τρόπο που δεν θα είναι μόνο κατευθυντήριε αρχέ, που είναι καλέ αλλά δεν αρκούν, γιατί αν θέλουμε να προχωρήσουμε ε, σε μια δεσμευτική συνθήκη μπορεί να μην εφαρμοστεί ποτέ ή να μην κυρωθεί ποτέ. Μπορεί δηλαδή να κερδίσουμε την πολιτική μάχη, αλλά όχι την αγώνα της εφαρμογής. Και αυτό είναι κρίμα. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε ταυτόχρονα και στα δύο παιδιά. Ευχαριστώ. Ναι, μακρηγόρησα, αλλά τι να κάνουμε. Ναι, είναι τεράστιο το θέμα, πράγματι. Θέλετε να πείτε δύο λόγια τέλος πολύ σύντομα, γιατί στις... Ε, ε, πρέπει να κλείσουμε στις 6 οι διερμηνείς ε, ε, τελειώνουν τη δουλειά τους, οπότε ένα λεπτό λοιπόν για να κλείσετε κι εσείς. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που μου ήρθαν στο μυαλό ακούγοντας τη συζήτηση για το, το ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης είναι εξαιρετικό να υπάρχει ένα κεφάλαιο μάλλον για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όμως αυτό θέτει τα όρια. Δηλαδή δεν επηρεάζει το υπόλοιπο της συμφωνίας. Για παράδειγμα, δεν λέει ότι όταν οργανώνετε την αγροτική σας οικονομία θα πρέπει να φροντίσετε τους μικρούς παραγωγούς. Η εμπορική πολιτική είναι η έκφραση των εμπορικών επιθετικών και αμυντικών συμφερόντων της Ένωσης. Αυτή είναι η ουσία της. Από εκεί και πέρα του υπάρχει ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη βεβαίω και συνεισφέρει και προς, προάγει κάποιες ιδέες, όμως δεν αρκεί. Έχουμε αυτή τη συζήτηση και πάλι σε σχέση με την Αφρική. Θα πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην, Αφρικα... Ε, στην Αφρική με τις απαιτήσει της, ενώ η Αφρική δεν είναι προετοιμασμένη, η κοινωνία των πολιτών δεν αναγνωρίζει τα ίδια ζητήματα, δεν υποστηρίζει τις ίδιες προτεραιότητες και έρχεται η Ευρώπη να επιβάλλει τις ε, απόψεις της και ίσως τα καταφέρει, αλλά αυτό δεν θα είναι καλό για την Αφρική. Με αυτή την ε, παρατήρηση νομίζω μπορούμε να κλείσουμε και τη συζήτηση. Θα ήθελα μήπως ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου να κάνει μια σύνοψη. Βεβαίω, λέει ο κύριο Λάνκε, δεν μπορούμε να ε, συνοψίσουμε όλη αυτή τη συζήτηση σε ένα λεπτό. Αλλά θα σταθώ σε αυτό που είπε ο συνάδελφο σωστά προηγουμένω. Έχει αλλάξει ο τόνο τη συζήτηση. Πριν από 10 χρόνια συζητάγαμε βέβαια για τον ΠΟΕ, για το περιβάλλον, για την βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά δεν ήταν στην κορυφή τη ημερήσια διάταξη. Αυτό σήμερα έχει αλλάξει. Επομένω, έρχεται η Μερικέ μερικές φορές με ρυθμούς αλληγκαριού, αλλά πρέπει να διαπιστώσουμε ότι έχουμε προοδεύσει. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ τη συντονίστρια, ευχαριστώ τους ομιλητές μας. Σας εύχομαι το καλύτερο. So, Karin, on 20... Σημείο 20. Κάριν, έχετε τίποτα στα διάφορα? Όχι. Ωραία. Η επόμενη μας συνεδρίαση στις 19 και 20 Φεβρουαρίου. Καλό απόγευμα.